Ich eröffne die heutige Sitzung. werde daran erinnern, dass ich immer pünktlich anfange. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι θα αρχίζουμε στην ώρα μας και σήμερα, αλλά και από εδώ και πέρα θα προσπαθήσω να είμαστε στην ώρα μας πάντα. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι και αυτή τη φορά μπορούμε να ξεκινήσουμε με διερμηνία σε όλες τις γλώσσες από σουηδικά, ιστονικά, μαλτέζικα, λιθουανικά και λετονικά ότι είμαστε συνδεδεμένοι και με το διαδίκτυο ότι η ημερήσια διάταξη μπορεί να θεωρηθεί εγκεκριμένη γιατί δεν βλέπω κανένα να ζητάει το λόγο και περνώ αμέσως στο σημείο 2. Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης. 2 με 3 Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι έχετε όλοι στο φακελό σας τα πρακτικά και σας ζητώ να ρίξετε μια ματιά και αν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης δεν μου πείτε ότι κάτι δεν είναι ορθό, θα θεωρήσω ότι εγκρίνονται τα πρακτικά της προηγούμενης ε, συνεδρίασης. Και περνάω στο σημείο 3. Έχω κάποιες πληροφορίες που θέλω να σας ε, παρουσιάσω. Στις 28 Σεπτεμβρίου, την προηγούμενη Δευτέρα δηλαδή, στο θέατρο Φλαζέ. Δεν ήμουν μόνη, ήταν κι άλλοι που είναι σήμερα παρόντες εδώ. Έλαβα χώρα στο, στην πρώτη τελετή απονομής βραβείων Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Λογοτεχνία, ήταν η Λιλερό, το πρόεδρος Μπαρόζο και 800 ονόματα από την ευρωπαϊκή πολιτιστική σκηνή. Ήταν μια εξαιρετική ε, τελετή και αυτό αυτό το βραβείο έχει σαν σκοπό να προωθήσει την πολυμορφία της λογοτεχνίας από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, 12 συγγραφείς παρόντες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 5.000 ευρώ είναι το βραβείο. Και υπάρχει κάθε φορά μια επιτροπή εθνική η οποία επιλέγει τους υποψήφιους. Αυτή τη φορά 12 χώρες ε, διόρισαν, ονόμασαν, επέλεξαν έναν συγγραφέα. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ε, εκδήλωση. Διαβάστηκαν και κάποια κομμάτια από τους ε, συγγραφείς αυτούς του χρόνου. 11 χώρες θα επιλεγούν θα του ζητηθεί δηλαδή να επιλέξουν ένα συγγραφέα και το 2011 άλλες 11 χώρες έτσι ώστε μέχρι σε τρία χρόνια 34 διαφορετικές επιλογές να βραβευθούν. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι και υποψήφιες χώρες. Και πρόκειται για το πολιτιστικό πρόγραμμα του 2007 και όλες οι χώρες που συμμετείχαν σε αυτό το πολιτιστικό πρόγραμμα το 2007 μπορούν να προτείνουν υποψήφιους. 34 χώρες λοιπόν. Επικεφαλής αυτής της Επιτροπής είναι ο γνωστός Henning Mankel. Εγώ πραγματικά γνωρίζω τον συγγραφέα αυτό, τον αγαπώ πολύ. Ξέρετε ότι έζησε τη μισή του ζωή στην Αφρική και μίλησε για την ευρωπαϊκή ταυτότητα, για τη σημασία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και συγκεκριμένα είπε ότι η Ευρώπη θα πρέπει πραγματικά να αρχίσει να δεσμεύεται στον πολιτισμό, ένα κεντρικό θέμα, και γιατί εάν δεν το κάνει μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένωση. Δεν υπάρχει ένωση χωρίς πολιτισμό και λογοτεχνία. Μας ευχαρίστησε λοιπόν για τις προσπάθειές μας και θα ήθελα επίσης να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποίησε την Biennale της Βενετίας για το βραβείο Λουξ. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι σας να κάνετε λίγη διαφήμιση για τα βραβεία και εδώ υπάρχει ένα βιβλιαράκι, μπορείτε να το πάρετε όλοι, που αναφέρεται στις τρεις ταινίες που επελέγησαν και έχει και μια μικρή παρουσίαση της συνέντευξης τύπου. Θα ήθελα να σας πω ότι στις 4 Νοεμβρίου θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να βλέπουμε τα έργα της ταινία. την εβδομάδα 3-4 Νοεμβρίου. Ή στις 3 ή στις 4 Νοεμβρίου, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω ακόμα ποια από τις δύο μέρες θα ξεκινήσει η προβολή. Οι τρεις σκηνοθέτες θα είναι παρόντες και θα τους ζητήσουμε να μας μιλήσουν για τα έργα τους, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, τι έχουν να πούν για την ε, ταινία που προετοίμασαν. Θα τους ζητήσουμε να έρθουν, να μας μιλήσουν, να αναφερθούν και στα πολύ σημαντικά θέματα που τους απασχόλησαν ο το πολιτικό άσυλο. Επίσης η αντιπροσωπεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα θέματα των εγκληματιών πολέμου και του ποινικού δικαστηρίου. Εμείς εδώ πραγματικά στην Επιτροπή Πολιτισμού πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά το θέμα αυτό και να κάνουμε διαφήμιση για αυτές τις προβολές ταινιών έτσι ώστε πολλοί συνάδελφοι να είναι παρόντες. Πρόκειται νομίζω για μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Σας δείχνω για άλλη μια φορά αυτή την μπροσούρα, αυτό το βιβλιαράκι, αλλά εγκαίρως θα σας ενημερώσουμε και πότε θα γίνει η προβολή των ταινιών. Θα είναι πάντα είτε το μεσημέρι, το απόγευμα ή ε, το βράδυ. Μετά δηλαδή το τέλος της συνεδρίασης ή το μεσημέρι την ώρα της ε, διακοπής. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να πάτε να δείτε αυτές τις ταινίε. Και τώρα προχωράω στο σημείο 4 τη ημερήσιας διάταξη, Έχουμε τον κύριο Ρόγκε εδώ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει μία μελέτη που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για τη νέα οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα. Όπως ξέρετε, έχουμε ήδη ξεκινήσει μια ολόκληρη μελέτη για την οδηγία αυτή και για τις νέες οδηγίες για τη διαφήμιση και υπήρξαν έντονες συζητήσεις, πολλοί ήταν υπέρ, πολλοί ήταν κατά. Και βεβαίως, όπως ξέρετε, η συζήτηση αυτή συνεχίζεται. Αυτό που πολλοί φοβόντουσαν, δεν ξέρουμε αν ήταν υπερβολικό. Είναι πολύ ενδιαφέρον πάντως το θέμα, συνεχίζει να προκαλεί έντονες συζητήσεις και είναι και ένα καλό παράδειγμα μελέτης, έρευνας που με πολύ πετυχημένο τρόπο έχει διεκπεραιωθεί. Ο κύριος Ρούγκε από το Kern European Affairs θα μας μιλήσει για λίγα λεπτά, δέκα λεπτά. Ξέρω ότι θα μπορέσει στο χρόνο που του έχουμε δώσει να μας παρουσιάσει το θέμα αυτό με ουσιαστικό και ε, πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθω εδώ και να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της έρευνάς μας εδώ στην Επιτροπή σας. Πολύ σύντομα θέλω να σας συστηθώ, να ξέρετε ποιοι είμαστε δηλαδή. Βασιζόμαστε εδώ στις Βρυξέλλες είναι η έδρα μας και γνωμοδοτούμε σε επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται με τα κοινωτικά όργανα αλλά και σε κυβερνητικά όργανα στα διάφορα κράτη-μέλη. Κυρίως ασχολούμαστε με θέματα πολιτισμού, δημιουργίας, μέσα ενημέρωση. Ε, καθορισμός πολιτικής κλπ. Πολύ σύντομα λοιπόν θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της έρευνάς μας όσον αφορά τους κανόνες που αφορούν τη διαφήμιση και όσον αφορά την οδηγία της ε, υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων. Νομίζω ότι δεν θα μου πάρει ούτε 20 λεπτά. Η μελέτη μας ε, λοιπόν επικεντρώνεται κυρίως στις τάσεις που υπάρχουν σήμερα όσον αφορά την κρίζα διαφήμιση, που είναι ένας νέος τρόπος διαφήμισης και που και η έρευνά παρουσιάζει τις τάσεις λοιπόν που υπάρχουν σε σχέση με την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Επίσης εξετάζει και τις επιπτώσεις που έχει η διαφήμιση στα παιδιά και κατά πόσο χρειάζεται και πώς προχωράει η αυτοδιαχείριση του θέματος αυτού στα διάφορα κράτη-μέλη. Κοιτάμε τις εξελίξεις έτσι όπως λαμβάνουν χώρα. Θα ξέρετε ότι η οδηγία δεν πρέπει να ενσωματωθεί παρά μόνο στα τέλη της χρονιάς θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτιση αυτή. Η γκρίζα διαφήμιση στα περισσότερα κράτη-μέλη δεν επιτρέπονταν μέχρι τώρα. Τα ελάχιστα λοιπόν στοιχεία που έχουμε όσον αφορά την κρίση διαφήμιση και τις επιπτώσεις που έχει στα έσοδα, τα έχουμε χρησιμοποιήσει. Καθορίζεται η γκρίζα διαφήμιση ως εξής. Είναι οποιοδήποτε τρόπος ο οποίος έχει να κάνει με οπτικοακουστική και εμπορική ανακοίνωση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ή ενός σήματος και περιλαμβάνεται σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Πρόκειται δηλαδή για διαφήμιση η οποία ουσιαστικά χώνεται μέσα στο πρόγραμμα χωρίς να είναι διαφήμιση αυτή καθ' αυτή. Η συζήτηση τα τελευταία χρόνια έχει γίνει για την κρίζα διαφήμιση και εντάσσεται στα πλαίσια της μείωσης των εσόδων από τις διαφημίσεις στα μέσα ενημέρωσης. Οι λόγοι είναι πολλοί. Η οικονομική κρίση βέβαια επί του παρόντος, η οποία όπως καταλαβαίνετε οδηγεί σε μείωση δαπανών από πλευρά του καταναλωτή, οπότε μείωση και των διαφημίσεων. Οφείλεται επίση στον κατακαιρματισμό του ακροτηρίου, γιατί όντω υπάρχουν νέα μέσα τεχνολογικά, διάφορε μέθοδοι για να αποφεύγουν τη διαφήμιση, για παράδειγμα, οι θεατέ κλπ. Η μείωση τώρα των εσόδων επηρεάζει φυσικά τον ε, τηλεοπτικό κλάδο. Σε πολλές χώρες τα έσοδα από τις διαφημίσεις είναι και η κύρια, ο κύριος παράγοντας που ενισχύει την τηλεοπτική παραγωγή. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, κάπου 60%. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, ορισμένοι θεώρησαν ότι η γκρίζα διαφήμιση μπορεί να είναι το μέσον για το μέλλον. Ιδιαίτερα ακριβώς τώρα που έχουμε αυτή την οδηγία. Αξιολογούμε λοιπόν το δυναμικό αυτό, τη δυνατότητα που υπάρχει μέσα από την κρίζα διαφήμιση επιτρέπεται ήδη και βέβαια προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε στοιχεία από συνομιλίες που έχουμε με τους καταναλωτές. Εμείς σας παρουσιάζουμε ε, την γκρίζα διαφήμιση ως μια νέα μορφή που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο. Όμως το κομμάτι της αγοράς που έχει η γκρίζα διαφήμιση στην τηλεόραση είναι βέβαια πολύ μικρό σε σχέση με την κανονική διαφήμιση. 2% το εκτιμάμε περίπου. Στα ευρωπαϊκά πλαίσια λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστούμε πώς θα προχωρήσουν τα έσοδα από την γκρίζα διαφήμιση. Ιδίως μάλιστα όταν σε ορισμένες χώρες δεν έχει επιτραπεί ακόμα. Το δυναμικό όμως είναι τεράστιο. Και η μελέτη παρουσιάζει διάφορα σενάρια. Από τις συζητήσεις που είχαμε καταλάβαμε ότι οι περισσότεροι διαφημιστές θέλουν την ελευθέρωση της γκρίζας διαφήμισης, την ε, επιτρέπεται δηλαδή, θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει μια νέα πηγή εσόδων. Και αυτό που εμείς πιστεύουμε και το κάνουμε και στη μελέτη μας είναι ότι εξηγούμε ότι η δυνατότητα αυτή ίσως να έχει υπερεκτιμηθεί κατά το παρελθόν και ίσως τελικά να αποτελέσει μια συμπληρωματική μόνο διαφήμισης. Τα επιχειρήματα τα εμφανίζουμε στη μελέτη μας, γιατί δηλαδή πιστεύουμε ότι θα πρόκειται για ένα μικρό συμπληρωματικό κομμάτι στην κανονική διαφήμιση. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν ελευθέρωσης της γκρίζας διαφήμισης, εξετάζουμε την κατάσταση όσον αφορά την οδηγία τώρα για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και πώς πάει εφαρμογείται στα διάφορα κράτη-μέλη. Κάναμε μία μελέτη σε όλες τις χώρες μέλη με συνεντεύξεις όπου ρωτάμε δύο πολύ απλά πράγματα. Πρώτον, αν η γκρίζα διαφήμιση επιτρέπεται στα κράτη-μέλη, θα επιτραπεί δηλαδή στα κράτη-μέλη και κάτω από ποια μορφή, και δεύτερον, κατά πόσο, υπάρχει, κατά πόσο αν υπάρχει εξαίρεση στην οδηγία, αυτή η εξαίρεση θα είναι σημαντική, γιατί υπάρχει ένα άρθρο που επιτρέπει να μην ενημερώνονται οι θεατές για το ότι πρόκειται για γκρίζα διαφήμιση. Στις αρχές του 2009 οι περισσότερες χώρες μέλη δεν είχαν ενσωματώσει ακόμα την οδηγία στην νομοθεσία τους. Όμως οι περισσότερες χώρες μέλη είχαν πει ότι σκόπευαν να επιτρέψουν την κρίζα διαφήμιση έτσι όπως προτείνεται από την οδηγία. Πολλές χώρες επίσης θέλουν να χρησιμοποιήσουν το άρθρο το οποίο επιτρέπει να μην ενημερώνονται οι τηλεθεατές για το ότι πρόκειται για γκρίζα διαφήμιση. Η Ρουμανία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Ιταλία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ισπανία και η Σουηδία. Υπάρχει λεπτομερής κατάλογος για τις θέσεις που έχουν υιοθετήσει τα διάφορα κράτη-μέλη, είναι στη διάθεσή σας εδώ. Σε ορισμένες χώρες έχει αλλάξει βέβαια τον τελευταίο μήνα η θέση των χωρών αυτών, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, που το εξετάζουν εκ νέου. Και σκοπεύουν να ξαναδούν την τελική εφαρμογή των κανόνων όσον αφορά την κρίζα διαφήμιση του χρόνου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν μας ζήτησε να εξετάσουμε τρία επιπλέον ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, για τις συνήθειες των παιδιών όσον αφορά τη τηλεόραση. Δεύτερον, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η διαφήμιση στην τηλεόραση πάνω στα παιδιά. Και τρίτον, θέματα που έχουν να κάνουν με την αυτορύθμιση. Πολύ σύντομα λοιπόν θέλω να θίξω αυτά τα τρία ζητήματα και μετά να ολοκληρώσω. Ο ορισμός του παιδιού πρώτα απ' όλα διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό βέβαια έχει σημαντικέ επιπτώσει, προκειμένου να μπορούμε να πούμε ότι ομοιογενώ εφαρμόζονται κανόνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ηλικία ενός παιδιού διαφέρει, όπως είπαμε, από χώρα σε χώρα. Ορισμένες δεν καθορίζουν καθόλου τα παιδιά σαν ομάδα απέναντι στη διαφήμιση. Ή δεν λένε τι εννοούν με το παιδικό πρόγραμμα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να έχουμε τις ίδιες προδιαγραφές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για την έρευνα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει σύγκριση. Δεύτερον, η μελέτη παρουσιάζει δεδομένα τα οποία δείχνουν την γενική συνένεση που υπάρχει μεταξύ των ερευνητών για το ότι η διαφήμιση επηρεάζει σε κάποιο βαθμό ε, τα παιδιά όταν αυτή περνάει στα μέσα ενημέρωσης και γι' αυτό και πολλοί είναι ιδιαίτερα σκεπτικιστές απέναντι στο θέμα της διαφήμισης γιατί δεν ενημερώνονται τα παιδιά για την διαφήμιση, τι σημαίνει ακριβώς είναι περίπου αναλφάβητη απέναντι στη διαφήμιση. Και γι' αυτό ρυθμίζεται πολύ αυστηρά η διαφήμιση που απευθύνεται σε παιδιά. Πολύ πιο αυστηρά από ότι η διαφήμιση για τους ανήλικες. Τα παιδιά κοιτάνε πολλά παιδικά προγράμματα. 69% των παιδιών κοιτάνε τηλεόραση και κατά την περίοδο που δεν έχει παιδικά προγράμματα. Τα παιδιά λοιπόν αποτελούν ένα στόχο για την διαφήμιση, πολλές φορές διαφήμιση που δεν προορίζεται για τα παιδιά. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας αυτό το γεγονός για να ρυθμίσουμε τις διαφημίσεις. Ο μέσος όρος που κοιτάνε παιδιά τηλεόραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται στην έρευνα. Στην κάτω χώρα 160 λεπτά την ημέρα. Αλλού 190, που είναι ακόμα πολύ χαμηλό αυτό το επίπεδο. Ενώ υπάρχουν χώρες όπως είναι η Αμερική και η Ιαπωνία, όπου τα παιδιά 4,5 ώρες την ημέρα κατά μέσο όρο βλέπουν τηλεόραση. Στην Ευρώπη 29 διαφημίσεις την ημέρα βλέπουν τα παιδιά. Το τελευταίο τώρα που θέλω να θίξω είναι το εξής μας ζήτησε το Κοινοβούλιο να κοιτάξουμε και τα θέματα της αυτορύθμισης. Το άρθρο 3α, τις οδηγίες που ζητάει από τα κράτη-μέλη να φροντίσουν να υπάρχει ένας κώδικας διοντολογίας όσον αφορά τις διαφημίσεις για παιδιά και να υπάρξει η προσέγγιση της αυτορύθμισης. Ο κύριος κώδικας διοντολογίας που αναφέρεται στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο όσον αφορά τη διαφήμιση έχει συζητηθεί και έχει προσαρμοστεί πρόσφατα στην Food and Beverage Communication. Περιλαμβάνει περισσότερες λοιπόν λεπτομέρειες τώρα. Και συμφώνησαν ενδιαφερόμενοι ότι ένα τέτοιο κώδικα δοντολογία μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό εφόσον σχεδιαστεί και εφαρμοστεί με ορθό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, η αποτελεσματικότητα βέβαια αυτών των κωδίκων όσον αφορά τη διαφήμιση που αποφθύνεται σε παιδιά μένει αποδειχτή, γιατί δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα οδηγία σε όλα τα κράτη-μέλη. Κοιτάξαμε επίση και τον αντίκτυπο τη διαφήμιση, πώ προχωράει. Είναι πολύ νωρίς βέβαια να πούμε πόσο σημαντική θα είναι η γκρίζα διαφήμιση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως πιστεύουμε ότι θα κρατήσει ένα μικρό κομμάτι της διαφήμισης στα οπτικοακουστικά μέσα. Και κατά πάσα πιθανότητα θα επιτραπεί στις περισσότερες χώρες μέλη. Και ότι η εξαίρεση θα ισχύει επίσης στα περισσότερα κράτη-μέλη μας ε, ζητήθηκε να προτείνουμε τομείς για παρέτερα έρευνα. Εμείς πιστεύουμε ότι όσον αφορά τις συνήθειες των καταναλωτών απέναντι στα οπτικοακουστικά μέσα, είναι κάτι που χρειάζεται, ιδίως για τα νεαρά παιδιά. Θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό όχι μόνο όσον αφορά τη διαφήμιση, αλλά και όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, για παράδειγμα, το copyright. Αν Πάντως το θέμα της γκρίζας διαφήμισης παραμένει καυτό, όπως είναι και τώρα. Πρέπει να δούμε και την προστατευσία που προσφέρει αυτή η γκρίζα διαφήμιση. Αυτό βέβαια αφού τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία. Ορισμένες χώρες, όπως η Ισπανία και η Αυστρία, ήδη έχουν αρχίσει να επιτρέπουν την γκρίζα διαφήμιση πριν ξεκινήσει η οδηγία. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η έννοια της... των αλφαβητισμού στη διαφήμιση θα μπορούσε να εισαχθεί και στην πρωτοβουλία της Επιτροπής που έχει κάτι αντίστοιχο για τα μέσα ενημέρωσης. Οπότε όσοι παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις θα μπορούν να στηρίξουν στα ευρωπαϊκά κοινωτικά όργανα παρετέρω τη σχετική ρύθμιση. Ευχαριστώ και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ρούγκε. Νομίζω ότι η τελευταία σας πρόταση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθότι το θέμα του κατά πόσο κατανοεί κανείς ε, το πώς λειτουργούν τα οπτικοακουστικά μέσα αυξάνει και τη δυνατότητα να αντιδράσει κανείς, να κατανοήσει ότι πρόκειται για διαφήμιση ή για ένα άλλο είδους μήνυμα. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό όχι μόνο σήμερα αλλά και τα επόμενα, ε, τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Μιλήσατε επίσης για αυτού του είδους την ε, διαφήμιση, την κρίζα διαφήμιση λέγοντας ότι μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον ε, έσοδο για τις διαφημιστικές εταιρείες. Βεβαίως, εάν η οδηγία προχωρήσει όπως ε, φαίνεται να κάνετε αυτή τη στιγμή τις προτάσεις σας, σαφώς και θα δημιουργηθούν νέες πηγές ε, εσόδων. Αλλά πρέπει να δούμε. Συνάδελφοι, θέλετε να κάνετε ερώτηση στον κύριο Ρούγκε. Η κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να μου δώσει κάποια στοιχεία όσον αφορά την γερμανική ορολογία. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι είναι ίσως νωρίς προς το παρόν για να μπούμε σε πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Σε πολλές χώρες, αλλά και στη Γερμανία, έχει ξεκινήσει ήδη η μεταφορά της οδηγίας αυτής στην εθνική νομοθεσία. Βέβαια, στην πράξη δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα προχωρήσει το θέμα αυτό και τι επιπτώσεις θα έχει, τι αντίκτυπο θα έχει. Η κυρία Πακ είπε και συμφωνώ μαζί της ότι και αυτοί που είναι υπέρ και αυτοί που είναι κατά αυτής της γκρίζας διαφήμισης, τοποθέτηση προϊόντων, έχουν κάνει προσπάθειες και μέσω των λόμπι και μέσω των ε, εσόδων που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν από αυτή τη δραστηριότητα Όλοι όμως συμφωνούν και οι υπέρμαχοι και αυτοί που είναι κατά ότι που δεν είναι λόγο δεν θα πρέπει να περιοριστούν εδώ τα μηνύματα και το εύρος των διαφημιστικών μηνυμάτων. Το θέμα τώρα είναι ποιοι είναι οι πραγματικοί αντίκτυποι, οι πραγματικές επιπτώσεις αυτών των ε, μηνυμάτων γκρίζας διαφήμισης και ότι πολλές φορές είπατε είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς αν πρόκειται για διαφήμιση ή για ένα άρθρο ή μια ε, ενημέρωση. Νομίζω ότι αυτή η σύγχυση είναι κάτι το οποίο κανείς δεν θέλει να αφήσει να περάσει. Ε, και θα ήθελα να ξέρω αν ο πολύ αυστηρός περιορισμός και έλεγχος ε, δεν θα οδηγήσει σε άλλου είδους αρνητικές επιπτώσεις. Το θέμα επίσης είναι αν μπορεί να υπάρξει αυτοέλεγχος. Τι πιστεύετε. Γιατί βεβαίως ε, ο αυτοέλεγχος στην οικονομία, στην κοινωνία είναι κάτι που δεν ξέρουμε αν μπορεί να έχει αποτελεσματικότητα. Ποια είναι η άποψή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ε, καλημέρα σας. Θα ήθελα να γνωρίζω αν μελετήσατε το ποσοστό που συνδέεται με τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων και με τις υπηρεσίες. Αυτό ε, προσεγγίζει και την ερώτηση της κυρίας Τρούπελ, δηλαδή σε σχέση με τα είδη προϊόντων που διαφημίζονται με αυτόν τον τρόπο και επιπλέον αν κάνετε διάκριση για τις δημόσιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, στη Γαλλία υπάρχουν διαφημιστικά μηνύματα που αφορούν ε, τα ταχυδρομεία, την κοινωνική ασφάλιση ή την υγεία. Και αυτό διαφέρει από μια διαφήμιση για το ποτό ή για το κάπνισμα. Έχετε δει λοιπόν τα ποσοστά. Κάνετε διάκριση στις μελέτες σας για τον αντίκτυπο αυτών των διαφημίσεων. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλε ερωτήσει. Κύριε Ρούγκε. Thank you very much. Uh, Σας ευχαριστώ. Σε σχέση με την πρώτη ερώτηση για τον αντίκτυπο και την ε, αξία της ε, διαφήμισης όπως παρουσιάζεται στην τηλεόραση δεν το εξετάσαμε αυτό. Εξετάσαμε το οικονομικό αντίκτυπο της γκρίζας διαφήμισης. Κάναμε προεκπολές από στοιχεία που είχαμε από αναλυτές της αγοράς μπορούμε να σας τις ε, δώσουμε αυτές τις προεκβολές, αλλά δεν κάναμε συγκεκριμένα προσέγγιση για την αξιολόγηση του κατά πόσο η γκρίζα διαφήμιση είναι κάτι επιθυμητό ή ανεπιθύμητο από την ε, άποψη της, ε, του περιεχομένου. Για το περιεχόμενο επίσης είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει διότι μέσα στο πεδίο της μελέτης ε, ήρθαμε σε επαφή με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, αυτούς που παριθμούνται στο παράρτημα της μελέτης και γενικά οι αντιδράσεις τους ήταν ότι οι κώδικες διοντολογίας, εάν ε, είναι καλά σχεδιασμένοι και εφαρμοσμένοι, μπορούν να είναι πολύτιμοι, αλλά όπως σας είπα νωρίτερα, είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε. Για την τελευταία ερώτηση, για τη διαφορά μεταξύ υπηρεσιών και προϊόντων, αυτό δεν το εξετάσαμε, γιατί για την ώρα η γκρίζα διαφήμιση δεν επιτρέπεται σε πολλά κράτη-μέλη. Και γι' αυτό είναι πολύ νωρί για να κάνουμε τέτοιου είδου αξιολόγηση. Αναφέρονται τα περισσότερο συχνά χρησιμοποιούμενα προϊόντα στην κρίζα διαφήμιση της ΕΠΑ Πρόκειται κυρίως για καταναλωτικά αγαθά και όχι για υπηρεσίε, και σίγουρα όχι για τις δημόσιες υπηρεσίε όπως αναφέρατε εσεί. αυτά για τι είπα. Σα ευχαριστώ. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό γιατί στα πλαίσια της νέας οδηγίας για τα οπτικοακουστικά μέσα και ο οικονομικός αντίκτυπος σε σχέση με τις διαφημίσεις είναι κάτι που μου δημιουργεί πρόβλημα. Εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ να δούμε και τον αντίκτυπο, παραδείγματο χάρη, στα παιδιά. Το περιεχόμενο, παραδείγματο χάρη, και αν αυτό σε σχέση με τα παιδιά και τους νέους έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε αν πραγματικά για την διαφημιστική αν θέλετε, αυτή η δραστηριότητα. Έχει υπολογιστεί ο αντίκτυπος για τα παιδιά και για τους νέους, ποιος είναι αυτός και πώς αντιμετωπίζεται από τους διαφημιστές. Συμφωνώ πολύ τους λέει η Πρόεδρος. Ποιος θα ήθελε το λόγο. Credo che ringrazio molto για questo. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση και συμμερίζομαι την παρέμβαση της συναδέλφου που μίλησε μόλις πριν από μένα. Θα ήταν πιστεύω πολύ ενδιαφέρον να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στα κεντρικά κίνητρα για τα οποία ε, έγινε η εμβάθυνση αυτή. Ζητήσαμε να κάνετε τη μελέτη αυτή για να δούμε ποια είναι, ποιος είναι ο αντίκτυπος στη συμπεριφορά των ανηλίκων πώς θα μπορέσουμε να βρούμε ισορροπία που θα πρέπει να τη βρούμε και που προβλέπεται και στην οδηγία. Πραγματικά μας τρομάζει το γεγονός γιατί είδαμε πως μόνο δύο έχουν μεταγράψει την ε, οδηγία και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στοιχεία που θα μας ε, λένε κατά πόσο η γκρίζα διαφήμιση που γίνεται συνήθως χωρίς ε, ειδοποίηση χωρίς ειδοποίηση για το γεγονός ότι είναι εξωτερικά προϊόντα σε σχέση με την παραγωγή κάθε φορά της, ε, του κάθε προγράμματος. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή αυτής της οδηγίας με μια πιο εις βάθος έρευνα για να δούμε ακριβώς ποιος είναι ο αντίκτυπος ε, αυτής της ε, γκρίζας διαφήμισης, στη συμπεριφορά ας πούμε ως προς τη βία, την κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών και το θέμα επίσης της ε, Ε, τυποποίησης της προσωπικότητας των ανηλίκων. Και αυτό σε σύγκριση με τα έσοδα που κάτι τέτοιο σημαίνει για τους ε, ε, παραγωγούς, για τα κανάλια. Να δούμε δηλαδή αν τα έσοδα αυτά μπορεί να αντιστοιχούν στο κοινωνικό κόστος που μπορεί να είναι και αυτό πολύ ψηλό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ μπορώ να συμφωνήσω με όλα όσα είπαν οι προηγούμενες ομιλήτρες. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Προς το παρόν η πρόταση που έχουμε για μένα δεν είναι επαρκής. Δεν ξέρουμε αυτού του είδους η κρυφή διαφήμιση, γιατί περί αυτού πρόκειται, τι επιπτώσεις έχει επί των νέων, επί των παιδιών. Πρόκειται πραγματικά για μία ύπουλη διαφήμιση, μία διαφήμιση η οποία δεν αναφέρεται σαν διαφήμιση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα αντιδράσουν τα κράτη-μέλη, ε, αν ναι ή όχι χρειάζεται σήμανση, αν υπάρχει ένας τρόπος, ε, εν πάση περιπτώσει, προειδοποίησης, γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι αν δεν εξετάσουμε ακριβώς τις επιπτώσεις και τον αντίκτυπο αυτής της κρυφής διαφήμισης, στα παιδιά και στους νέους μπορεί να υπάρξει πάρα πολύ σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά και επιπτώσεις ε, τις οποίες σήμερα δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε. Γι' αυτό και θα ήθελα εγώ, ε, ενώ ακόμα δεν έχει μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες αυτή η οδηγία, να εξετάσουμε αυτές τις επιπτώσεις πριν προχωρήσουμε ε, στην εφαρμογή και στην υλοποίηση. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ζητήσαμε σήμερα αυτήν την μελέτη διαφήμιση και ανήλικη είναι το θέμα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε το θέμα. Ακούσαμε κάποιες πρώτες εκτιμήσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις. Αυτό που μας αφορά ιδιαίτερα είναι ο αντίκτυπος επί των νέων. Ίσως ε, τα θέματα δεν έχουν ακόμα εξεταστεί αρκετά ώστε να γίνει μια πλήρης παρουσίαση. Ε, σίγουρα το θέμα δεν το έχουμε εξαντλήσει. Λυπάμαι. Ε, και εγώ δεν ήξερα ποιο ήταν το περιεχόμενο αυτής της μελέτης και ζητώ συγγνώμη γιατί άλλο είναι ο τίτλος του θέματος και άλλο το περιεχόμενο που ακούσαμε τουλάχιστον. Κύριε Ρουγκέ, έχετε το λόγο. Να κάνω μια σύντομη παρατήρηση. Όπως μας ανατέθηκε η μελέτη, ήταν μια σύντομη μελέτη και ήταν μάλλον μια προμελέτη, προκειμένου να εντοπίσει νέους τομείς έρευνας. Και αν δείτε τα συμπεράσματα της μελέτης, θα δείτε ότι εκεί εξετάζουμε αυτά που μόλις αναφέρετε και προτείνουμε να υπάρξουν νέε έρευνες πάνω σε αυτού του τομεί. Δηλαδή εμεί δεν καταλήγουμε σε μια τελική σύσταση όσον αφορά, ή τελικό συμπέρασμα όσον αφορά τι επιπτώσεις της ε, κρίζα αυτής διαφήμιση πάνω στα παιδιά. Λέμε ότι πρέπει εντοπίζοντα νέους τομείς να ερευνήσουμε παρετέρω. Το καταλάβαμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε για αυτό που μας παρουσιάσατε και επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται περαιτέρω εγγρασία. Εμείς θα δούμε τι ακριβώς απόφαση θα πάρουμε, τι θα κάνει το Κοινοβούλιο και με ποιο τρόπο θα το κάνει. Σας ευχαριστούμε ε, πολύ πάντως για την παρουσίασή σας και ζητώ συγγνώμη γιατί δεν είχαμε μια οθόνη ε, με την οποία θα μας παρουσιάζατε κάποιες διαφάνειες. Και περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Σήμερα έχουμε από το Εδώ έχουμε τρία άτομα από το Policy Department. Ξέρετε ότι ο σκοπός του είναι να μας διευκολύνουν, να μας ελαφρύνουν, αν θέλετε, λίγο τη καθημερινή μας ζωή. Ο κύριος Ολιβάρης Μαρτίνες, ο οποίος είναι υπεύθυνος για πέντε επιτροπές και ο οποίος θα μας κάνει και μια μικρή εισαγωγική ε, παρουσίαση και κατόπιν θα δώσουμε και στις δύο κυρίες το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται να παρουσιάσουμε την υπηρεσία μας, την υπηρεσία ερευνών και το τμήμα αυτό που ασχολείται με την εκπόνηση πολιτικών μελετών. Ε, θέλουμε να ενημερώσουμε τους νέους κυρίως βουλευτές ότι το 2004 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναδιορθώσει τις υπηρεσίες αρρωγής προς τους ευρωβουλευτές έτσι ώστε να συμπεριλάβει και τις μονάδες έρευνας που μέχρι τότε δούλευαν στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και να τις συμπεριλάβει στην ίδια τη δομή άμεση στήριξη, άμεση αρρωγή προ τους ευρωβουλευτέ. Δηλαδή, τις γενικές, ε, τη Γενική Διεύθυνση, λοιπόν, πόλη για τι εσωτερικέ και εξωτερικέ πολιτικές Είναι μια μονάδα έρευνας η οποία δουλεύει πολύ στενά με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και έχει ως στόχο να παρουσιάσει πραγματογνωμοσύνη που εσείς θεωρείτε ότι σας είναι χρήσιμη για να επιτελέσετε το έργο σας. Δεν είναι μια ατομική υπηρεσία, αλλά στηρίζουμε τις κοινοβουλευτικές εργασίες των κοινοβουλευτικών ε, οργάνων. Όλο και περισσότερε δυσκολίε αντιμετωπίζουν οι ευρωβουλευτές επειδή τα θέματα είναι ιδιαίτερα περίπλοκα, επειδή οι νομοθετικές διαδικασίες είναι περίπλοκες. Έτσι λοιπόν, για να έχουμε καλύτερη ρύθμιση, που είναι βασικό στόχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στο νομοθετικό του έργο το Κοινοβούλιο, θεωρήσαμε χρήσιμο να προσφέρουμε στις κοινοβουλευτικέ ε, ε, επιτροπές τις γνώσεις μας και να μπορούμε και να προσφύγουμε και εκτός κοινοβουλίου σε άλλους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που μπορούν να μας βοηθήσουν όπως έγινε και σήμερα που ακούσαμε τα αποτελέσματα έρευνας που ανατέθηκε σε εμπειρογνώμονες εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν και οι έρευνες που γίνονται από μάς και εκείνες που γίνονται εκτός Κοινοβουλίου είναι υπό την ευθύνη των θεματικών μονάδων που στηρίζουν τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Η μονάδα Β υπό την κυρία Ολιβέηρα είναι αυτή που συνεργάζεται άμεσα με την ομάδα άμεσης στήριξης προς τους ευρωβουλευτές. Ο κύριος Στίβεν Σόλτερ είναι επικεφαλής. Δεν χρειάζεται να σας υπογραμμίσω ότι οι υπάλληλοι που κάνουν αυτή τη δουλειά είναι άνθρωποι με πολλές γνώσεις που γνωρίζουν με κάθε λεπτομέρεια την κοινοτική πολιτική. Όμως δεν είναι εμπειρογνώμονες για όλα τα θέματα. Καμιά φορά μπορεί να απευθυνθούμε στο Ινστιτούτο Παστέρ, για παράδειγμα, για να ενημερωθούμε για κάποιο, κάποια θέματα ή αλλού. Οι συνάδελφοι αυτοί που είναι οι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ειδικοί στον εντοπισμό των ε, θεμάτων. Παρακολουθούν τη ζωή των κοινοβουλευτικών επιτροπών σε καθημερινή βάση, γνωρίζουν πώς δουλεύουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ε, γνώσεις που μας έρχονται απ' έξω. Ως διευθυντής εγώ είμαι υπεύθυνο καταρχήν για το συντονισμό μεταξύ της γραμματείας των κοινοβουλευτικών ε, επιτροπών και των θεματικών τμήματων. Τα οποία θεματικά τμήματα δίνουν πληροφορίες, κάνουν την έρευνα και τη στήριξη που, που χρειάζεται για τις κοινοβουλευτικές εργασίες. Ένα μικρό σχόλιο θέλω να κάνω εδώ, κυρίως για τους νέους ευρωβουλευτές που ξεκινάνε φέτος με τη θητή αυτή. Θέλω να σας πω ότι οι μελέτες που γίνονται, οι έρευνες τόσο στο εσωτερικό όσο και εκτός κοινοβουλίου αποτελούν ένα μέσο που έχετε στη διάθεσή σας, που είναι στην υπηρεσία σας. Τη χρησιμότητά του, την ισχύ του, αυτό το κρίνετε εσείς θεσμικά και πολιτικά αποφασίζετε πάνω σε αυτό. Εμείς σας δίνουμε τις πληροφορίες και εσείς τις χρησιμοποιείτε όπως πιστεύετε ότι μπορούν να σας φανούν χρήσιμες για τις εργασίες σας. Καμία μελέτη δηλαδή που κάνουμε εμείς, καμία έρευνα δεν αντικαθιστά τον πολιτικό διάλογο που γίνεται μέσα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Εννοείται αυτό. Συνεπώς, εσείς έχετε την ευθύνη να εντοπίζετε τη θεσμική αναγκαιότητα για να ζητήσετε μελέτες και να μας πείτε ποιο θέλετε να είναι το περιεχόμενό τους. Είναι επίσης αρμοδιότητα της δικιάς σας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να δει πώς θα χρησιμοποιήσει σε θεσμικό επίπεδο την μελέτη που θα σας προσφέρουμε εμείς. Η Γενική Γραμματεία, από την άλλη, διασφαλίζει την ποιότητα και την πολιτική αυτονομία, ανεξαρτησία των μελετών αυτών, ουδετερότητα. Εγώ ως διευθυντής, από τη μια όπως σας είπα συντονίζω τις εργασίες, από την άλλη μεριά είμαι υπεύθυνο για τα οικονομικά. Εγώ δηλαδή ε, φροντίζω για τους πόρους προκειμένου να ζητήσουμε έρευνες, κάνουμε διαγωνισμό βέβαια και εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη Στήριξη των οικονομικών συμφερόντων της ε, κοινότητας. Τώρα, κυρία Πρόεδρε, προτείνω να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κονζάλο Μασέντου, ο οποίος εκ μέρους των θεματικών τμήματων θα σας παρουσιάσει περισσότερο σε λεπτομέρειες πώς συνεργαζόμαστε με διάφορες συμβουλευτικές εταιρείες που κυρίως έχουν έδρα τους στις Βρυξέλλες. Το σημαντικό που θα πρέπει να γνωρίζετε για τη δομή μας είναι ότι βρισκόμαστε στην ίδια δομή όπως και η γραμματεία της Επιτροπής ε, Πολιτισμού, δηλαδή ο κ. Ολιβέρας, ε, είναι ο διευθυντής μας, γνωριζόμαστε και συζητάμε τις εργασίες της Επιτροπής μαζί τους επί τη βάση των δικών σας ετοιμάτων φυσικά. Τώρα, όσον αφορά τη δική μας ε, ε, ισχύ ιδιαιτερότητα, ε, αυτή είναι ότι κυρίως εργαζόμαστε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής. Υπάρχουν πολλοί εμπειρογνώμονες, πολλές μελέτες εκτός Κοινοβουλίου, αλλά το ερευνητικό αίτημα μια Επιτροπής βασίζεται σε κάτι συγκεκριμένο που γίνεται σε κινητικό επίπεδο και μπορείτε εσείς να φτιάξετε την εντολή, τις απαιτήσει για μια μελέτη. Δεύτερο πλεονέκτημα του τμήματός μας είναι ότι εργαζόμαστε με ένα κάποιο βαθμό αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας από τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, γιατί είμαστε εντός της διοίκησης του Κοινοβουλίου και επίσης συνεργαζόμαστε Μάλλον ε, είμαστε ανεξάρτητοι και από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο, αλλά και ανεξάρτητοι από τι ε, μυριάδε ε, ομάδων πίεση που εδράζονται και λειτουργούν στι Βρυξέλλε και προσπαθούν να επηρεάζουν τα αποτελέσματα των ερευνών. Το άλλο πλεονέκτημα που σα ανέφερα είναι ότι εργαζόμαστε στην ίδια Γενική Διεύθυνση όπω και η Γραμματεία τη Επιτροπή Πολιτισμού και γι' αυτό και είμαστε σε θέση εύκολα να συζητήσουμε μαζί του εκ των προτέρων ποια είναι τα ενδιαφέροντα της Επιτροπής στους επόμενους μήνες, ώστε να προγραμματίσουμε τις εργασίες μας. Η μία έκθεση με τον, για την οποία εργάζεστε είναι ο διάλογος ε, ε, μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρηματικού κόσμου ε, που, θα, που έχει ήδη αρχίσει να μελετάτε στην Επιτροπή και έτσι μπορούμε να κάνουμε έρευνες που θα φτάσουν έγκαιρα σε εσά όταν οι εκθέσεις αυτές συντάσσονται. Ο πρώτος λοιπόν προγραμματισμός είναι πολύ σημαντικός. Στόχος ε, μας ως ακροατήριο είναι η Επιτροπή αυτή, αλλά έχουμε και άλλα σώματα στο Κοινοβούλιο για τα οποία εργαζόμαστε μετά από έτοιμα του Προέδρου ή των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών και ίσως και των γενικών διευθύνσεων και των διευθυντών. Τώρα, Όσον αφορά τον προπολογισμό, χονδρικά ήταν 240.000 ευρώ πέρυσι, λίγο λιγότερο από ό,τι ήθιστε, γιατί ήταν εκλογικό έτος. Υπήρχαν πολύ, υπήρχε πολύ λίγη κοινοβουλευτική εργασία στα μέσα του έτους, πράγμα το οποίο επηρεάζει το πώς μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε τον προπολογισμό. Εμεί θα ταπανίσαμε τι 230.000, δηλαδή τα περισσότερα χρήματα για φέτο. η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών στην Σύνοδο του Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο αποφάσισε να δώσει σε όλες τις επιτροπές ένα νέο προπολογισμό. Περίπου 50.000 ευρώ θα δοθούν στην Επιτροπή Προπολογισμού και εδώ σας στρογγυλοποιώ κάπως τα νούμερα. Όσον αφορά την εξέλιξη του προπολογισμού, σταδιακά αυξάνεται από τότε που δημιουργήθηκε το τμήμα μας το 2004. Τότε ήταν συμβολικό το ποσό, ήταν λιγότερο από 50.000 ευρώ. Τώρα έχουμε φτάσει στα 300, στις 350.000 ευρώ ετησίω περίπου. Αυτό ισχύσει για το 2008 και πιθανότατα αυτό θα είναι και ο προπολογισμό για το 2010. Εν περιπτώσει κάπω σε αυτή την τάξη μεγέθου Σε αυτή τη διαφάνεια στόχο έχουμε να σας δώσουμε να σας δείξουμε ότι εργαζόμαστε εσωτερικά αλλά και εξωτερικά με εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη. Ε, συνήθως συντάσσουμε εκθέσεις μέσω σημειωμάτων και συνοψίζουμε έτσι την κατάσταση. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες μπορεί να είναι προφανείς για τα παλιά μέλη ε, της Επιτροπής, υπάρχουν όμως και πολλά νέα μέλη σε αυτή την Επιτροπή. Όταν κανείς θέλει να υποβάλει ένα αίτημα στην Επιτροπή ε, πολιτισμού και σε όλες τις επιτροπές πάντοτε αυτό γίνεται στις συνεδριάσεις των συντονιστών. Δηλαδή, οποιοδήποτε βουλευτής ε, διαφέρει για κάποια μελέτη θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον συντονιστή του για να υποβάλει το θέμα και να μπει αυτό στην ημερήσια διάταξη. Διότι η τελική απόφαση λαμβάνεται σε αυτήν την επιτροπή, ε, στη συνάντηση μάλλον. Επειδή η Επιτροπή Πολιτισμού συνεδριάζει από καιρούς καιρών, ορισμένες επιτροπές έχουν ε, ετοιμάσει έναν άλλο τρόπο για να να στέλνουν αυτέ οι μελέτε ή σημειώσετε. Μέσω γραπτική διαδικασία όχι συντονιστέ, μέσω ή οι μέσω γραπτής διαδικασια όπου οι συντονιστέ μέσω email συνεννοούνται. Μέχρι στιγμή στην Επιτροπή Πολιτισμού δεν έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον αν χρειαστεί. Αυτά είναι τα βασικά ερευνητικά εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας, οι μελέτες, είναι αυτό το είδος εγγράφου που λάβατε σήμερα, ανάμεσα στα έγγραφα που λάβατε και που σας παρουσιάστηκε νωρίτερα. ένα σημείωμα είναι κάτι συντομότερο που δίνει σύντομες πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα. Και υπάρχει άλλο ένα εργαλείο που μπορεί να είναι χρήσιμο εδώ και έχει χρησιμοποιηθεί πολύ σε άλλες επιτροπές, εδώ όχι ακόμα. Και ονομάζεται εργαστήριο. Είναι παρόμοιο με μια ακρόαση με την έννοια ότι διάφοροι εμπειρογνώμονες καλούνται να μιλήσουν για ένα συγκεκριμένο θέμα αλλά διοργανώνεται από εμά στην Επιτροπή Μελετών, από το Τμήμα μάλλον Μελετών, ακολουθούμε διαφορετικού κανόνε. Ε, Εμεί αναζητούμε δηλαδή του εμπειρογνώμονε και χρησιμοποιούμε τον προπολογισμό μα για να του καλέσουμε. Μπορεί να υπάρχουν δύο τύπων ε, σεμινάρια. Μη μία σειρά ανθρώπων μιλούν για, διάφορα θέμα, για κάποιο θέμα και προσπαθούν να διαφωτίσουν ένα περίπλοκο θέμα, επί το οποίο καθένα από αυτού που έχουν προσκληθεί είναι εμπειρογνώμονε ή μπορεί να υπάρχει ένα πιο αντιφατικό εργαστήριο όπου ακούγονται διαφορετικές απόψεις για το ίδιο θέμα. Τώρα, ε, υπάρχουν και συγκεκριμένα δελτία με πληροφορίες που υπάρχουν για όλους τους τομείς πολιτικής και αυτά είναι δημοσιευμένα στο ίντερνετ. Εδώ συνοψίζουμε την εργασία μας, θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη, αξιόπιστη και κέρια. Δηλαδή η γλώσσα που χρησιμοποιείται να είναι καθαπλή, καθημερινή γλώσσα, αυτή που χρησιμοποιείται στην πολιτική συζήτηση, αξιόπιστη με την έννοια ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται εκεί να είναι σωστά και βέβαια οι πολιτικοί θα τα ερμηνεύσουν και κέρια ε, με την έννοια ότι η μελέτη αυτή θα πρέπει να είναι σχετική με το έργο της Επιτροπής και όχι με τα πολλά και διάφορα θέματα που μπορεί να θεωρηθούν ε, πολιτισμός, ε, παιδεία ή πολιτική για τα οπτικοακουστικά. Να είναι ένα εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει τους βουλευτές στην εργασία τους σε αυτή την Επιτροπή. Σας παρουσιάζουμε τις αρχές που διέπουν την εργασία μας. Δεν πρόκειται για δική μας εφεύρεση. Οι περισσότερες από αυτές τις αρχές συμπεριλαμβάνονται και στον ε, δημοσιονομικό κανονισμό. Είναι, ο νόμος είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία επί της οποίας εργαζόμαστε, επί της οποίας βασιζόμαστε όταν ε, κάνουμε ε, πρόσκληση για υποβολή προσφορών, Ακεραιότητα, αυτό είναι κοινή λογική, Αυτό σημαίνει ότι όποτε ξεκινά μία διαδικασία για εξωτερική πραγματογνωμοσύνη, γίνεται μια συγκεκριμένη επιτροπή, εξετάζει τις ε, δυναμίες και τα ε, δυνατά στοιχεία κάθε προσφοράς και αιτιολογεί την επιλογή της. Ε, το τελευταίο στοιχείο είναι η λογοδοσία. Λογοδοσία στην ίδια την Επιτροπή. Δηλαδή θέλουμε να σας ε, ενημερώνουμε για το τι κάνουμε, δεν θέλουμε να είμαστε ένα απομονωμένο ερευνητικό τμήμα το οποίο θα εμφανίζεται μία φορά το χρόνο. Ο κ. Ε, Ολιβάρης τακτικά ε, απευθύνεται στην πρόεδρο της Επιτροπής, στην κυρία Πάτκα, της γνωστοποιείται ότι έχουμε κάνει, τι μελέτες έχουμε κάνει κτλ. Και στα έγγραφα που παίρνετε από ότι γραμματεία για τις συνεχιζόμενες εργασίες της Επιτροπής υπάρχει πάντοτε ένα τμήμα των μελετών που αφορά ένα, ένα κεφάλαιο μάλλον που αφορά τις μελέτες, σε, σε ποιο στάδιο βρίσκονται, πότε θα ολοκληρωθούν κτλ. Examples of what we're working on at the moment. I've already mentioned the University Business Dialogue. Εδώ έχουμε ένα τμήμα για τις τρέχουσες μελέτες, ε, ας πούμε αυτή που αφορά το διάλογο μεταξύ των πανεπιστημίων και του επιχειρηματικού κόσμου, την μεταρρύθμιση της πολιτικής για την νεολαία, την ανακοίνωση για τις την εκπομπές, πρόγραμμα Εράσμου και εφαρμογή τη ε, σύμβασης τη UNESCO. Όλα αυτά αποφασίστηκαν από του συντονιστέ τον Ιανουάριο του 2009. Είναι το πρόγραμμα εργασία τη Επιτροπή. Άλλη βασική εργασία που κάναμε πρόσφατα ήταν το πρακτικός οδηγός. Σας έχει διανεμηθεί σήμερα ένα μικρό κίτρινος οδηγός. Όχι, αυτός είναι ο γκρι οδηγός που έχετε, ο κίτρινος. Είναι μια εισαγωγή στην κοινοβουλευτική εργασία μιλάει για τις βασικές, τη βασική δουλειά της Επιτροπής στην τελευταία θητεία και το τι προβλέπεται για αυτήν τη θητεία. Να σας δείξω και πού μπορείτε να βρείτε τα έγγραφά μας. Το site του ίντερνετ. Να σας πω ότι η έρευνα που γίνεται για αυτή την επιτροπή βασικά δημοσιεύεται στο ίντερνετ. Σχεδόν τα πάντα δημοσιεύονται στο ίντερνετ και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έχουμε και ένα δελτίο τύπου, ένα newsletter ε, που εκδίδεται μηνιαία και δίνει πληροφορίες για τις τελευταίες μελέτες και ε, σημειώματα τα οποία έχουμε ολοκληρώσει. Εδώ έχετε την λίστα με τα ονόματα. Είμαστε και οι τέσσερις μας εδώ σήμερα και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πάρα πολύ αξιόλογη εργασία για μας, τους πιο παλιούς. Ξέρουμε πολύ καλά πού μπορούμε να στραφούμε όταν ψάχνουμε κάτι, ποιο είναι η πηγή, τι υπάρχει, τι είναι διαθέσιμο και πραγματικά Χρησιμοποιώντας το ίντερνετ βλέπουμε ότι τα περισσότερα στοιχεία υπάρχουν και αυτό είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμο και αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Η κυρία Τρίπουλα έχει ζητήσει το λόγο. Δεν θα ήθελα όμως να συζητήσουμε για το θέμα αυτό πολύ ώρα, γιατί η κυρία Κοντά είναι ήδη εδώ. Σας ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση μόνο. Καταρχήν, ε, ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση. Στο σημείο 3, όταν αναφερθήκατε στις, στα δυνατά σας σημεία, είπατε ότι μπορείτε να κινητοποιήσετε εμπειρογνώμονες, καθηγητές, ακαδημαϊκούς και μιλήσατε επίσης για τους διαγωνισμούς και την υποβολή προτάσεων. Θα ήθελα να ξέρω, εδώ η οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα ανήκει στο δικό σας τομέα. Φαντάζομαι ναι και πριν λίγο έγινε μια παρουσίαση η οποία καθόλου δεν μας ικανοποίησε. Και θα πάρω σαν παράδειγμα αυτή την τελευταία παρουσίαση. Πώς διαλέξατε το think tank ή τους καθηγητές ή τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα κάνουν αυτή την παρουσίαση. Γιατί αν πραγματικά πάρουμε αυτό το τελευταίο παράδειγμα της παρουσίασης που δεν μας ικανοποίησε, Πώς μπορούμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Στη σελίδα 23 αυτού του εγγράφου θα δεις και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Μα ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημά μου. Ζητάμε μία μελέτη. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που είδαμε σήμερα. Θα ήθελα να ξέρω, να καταλάβω πώς μπορούμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον, δίνοντας πολύ πιο συγκεκριμένες οδηγίες και εντολή. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, λέει η Πρόεδρος, ο κύριος Ολιβέρας μπορεί να απαντήσει. Ποιος από τους κυρίους ή κυρίες παρόντες εδώ θα ήθελε να απαντήσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγκεκριμένα όταν αφορά το θέμα μας εξωτερικές μελέτες, μελέτες που γίνονται από εξωτερικούς ε, εμπειρογνώμονες, η διαδικασία είναι η εξής. Πάντα κάνουμε ανοιχτούς διαγωνισμούς και βεβαίως τηρούμε πάντα τον ε, ε, κανονισμό, ο δημοσιονομικός κανονισμός είναι εδώ Ευαγγέλιο για μας. Πάντα όμως, πριν κάνουμε κάτι τέτοιο, προσπαθούμε να βρούμε ε, εμπειρογνώμονες στο εσωτερικό της ε, υπηρεσίας. Όπως σας είπα όμως για τον πολιτισμό, ο κύριος Μασέντο και η κυρία Μαρία Κουνεντέιντο που είναι εδώ, η οποία είναι εμπειρογνώμονας και όχι υπάλληλο. Δεν έχουμε άλλο προσωπικό. Όταν πρόκειται λοιπόν για μια μελέτη η οποία βρίσκεται στην κατηγορία των μελετών κάτω από 60.000, προσπαθούμε στο εσωτερικό των κρατών μελών να βρούμε 20 τουλάχιστον Ινστιτούτα, πανεπιστήμια. Έχουμε ένα κατάλογο κάνουμε μια προηγούμενη προμελέτη, αν θέλετε, για να εντοπίσουμε τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν αυτήν την ε, μελέτη. Όταν ξεπερνάμε το ποσό των 60.000, δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα ο διαγωνισμός. Δεν είναι όμως αυτό η περίπτωση της προηγούμενης μελέτης που σας παρουσιάστηκε σήμερα. Όταν γίνεται επίσημη δημοσίευση υπάρχει μια προθεσμία και δίνεται μια σύμβαση πλαίσιο. Στη σημερινή σας παρουσίαση, την οποία μόλις ακούσατε, υπήρξε σύμβαση πλαίσιο σε έναν εμπειρογνώμονα, σε έναν ειδικό, ο οποίος μέχρι τώρα είχε κάνει πολλές μελέτες οι οποίες ικανοποίησαν την Επιτροπή σας. Όσον αφορά τις ε, τεχνικές, ε, αν θέλετε, προϋποθέσεις, πρέπει να σας πω ότι οι επιδόσεις ήταν ικανοποιητικές. Από εκεί και πέρα, σήμερα ακούσατε μια πρώτη παρουσίαση, μια προμελέτη μελετη όπως σας είπε ε, και ο κύριος που έκανε την παρουσίαση και βεβαίως εσείς θα αποφασίσετε αν ναι ή όχι θα συνεχίσετε την μελέτη περαιτέρω. Πρόεδρος. Κατάλαβα. Από εδώ και πέρα εμείς λοιπόν αποφασίζουμε αν θα συνεχίσουμε και με ποιο θέμα θα συνεχίσουμε και αν θα συνεχίσουμε με αυτούς ή με κάποιους άλλους. Επιτρέψτε μου, κυρία Πρόεδρε, να σας πω ότι οι μελέτες αυτές, οι έρευνες αυτές είναι πρωτοβουλία κάποιων επιτροπών ή κάποιων μελών του Κοινοβουλίου. Από τη στιγμή που το θέμα εγκρίνεται, αν θέλετε, από μέρους των συντονιστών, η μελέτη γίνεται μελέτη της Επιτροπής. Την προηγούμενη θητεία υπήρξαν κάποιες παρεξηγήσεις, παρανοήσεις. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η μελέτη είναι μελέτη της Επιτροπής και πάντα δημοσιεύεται. Η κυρία Κοντά είναι εδώ. Πολύ σύντομα λοιπόν με τις ερωτήσεις σας παρακαλώ πολύ. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς οι οποίοι μας έκαναν τις παρουσιάσεις. Ήταν πολύ ε, ενδιαφέρουσες. Όσον αφορά την γκρίζα διαφήμιση, ακούσαμε πολύ κριτική. Όσον αφορά όμως το περιεχόμενο και από τη στιγμή που δεν έχει μεταφερθεί η οδηγία αυτή στην νομοθεσία των κρατών μελών, δεν μπορώ να καταλάβω τι περαιτέρω ε, ανάλυση μπορούμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γραφτεί στα πρακτικά. Ακούσαμε έντονη κριτική αλλά κοιτάξτε πραγματικά πώς έχουν τα πράγματα. Για μένα ήταν χρήσιμη η παρουσίαση που ακούσαμε. Euh, non, je voulais euh, dire simplement deux Euh, Θέλω να αναφερθώ λίγο στην προηγούμενη θητεία που δύο φορές ήμουν πρόεδρος επιτροπής και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι πρώτον το θεματικό τμήμα είναι πάρα πολύ χρήσιμο πραγματικά αλλά υπό μία προϋπόθεση και σήμερα φάνηκε αυτό ότι δηλαδή οι ευρωβουλευτές και συνεπώς οι ίδιοι συντονιστές θα πρέπει να ξέρουν με ακρίβεια πού θα επικεντρωθεί η μελέτη. Δεν θέλω να κρίνω τώρα τη ποιότητα της σημερινής παρουσίασης. Νομίζω ότι δεν έφταιγε η παρουσίαση, ότι έφταιγε ο στόχος, ότι δηλαδή το θέμα δεν είχε καθοριστεί συγκεκριμένα. Γιατί αν πρόκειται για τέτοιες επιπτώσεις, γκρίζας, διθύμψης κτλ. δεν θα έπρεπε να απευθυνθούμε και στον ιατρικό κόσμο, στην ψυχολογία. Γιατί το ξέρουμε ανέκαθεν ότι η γκρίζα διαφήμιση οικονομικά προσθέτει ότι δεν είναι η βάση. Η διαφήμιση εξακολουθεί να υπάρχει, εννοείται. Αν διαβάσουμε αυτά που λένε επαγγελματίε σοβαρά, το βλέπουμε. Αλλά πολύ σωστά πάντως είπαν όσοι μίλησαν πριν από μένα ότι πρέπει να ξέρουμε πού επικεντρωνόμαστε. Γιατί να υπάρχουν χώρες και χώρες για τις οποίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξέρουν τις επιπτώσεις που έχει η γκρίζα διαφήμιση, αλλά να ακούσουν τη γνώμη του ιατρικού κόσμου. Συνεπώς, η θυματική μονάδα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, εφόσον εμείς ξέρουμε τι θέλουμε ακριβώς. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η διευκρίνηση. Να θέτουμε σωστές ερωτήσεις για να παίρνουμε σωστές απαντήσεις τη σωστή στιγμή. Ευχαριστώ πολύ στο τμήμα εκπόνησης μελετών και ελπίζω και στο μέλλον να συνεχιστεί η συνεργασία μας, εμείς να θέτουμε τις σωστές ερωτήσεις και εσείς να βρίσκετε τους καλούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες για να μας δίνουν τις καλές απαντήσεις. Η κυρία Οντιλ Κοντά είναι εδώ. Θέλω να την χαιρετήσω. Είναι η Γενική Διευθύντρια της, του Τμήματος Παιδείας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αν θέλετε μετά την Επίτροπο το πιο σημαντικό άτομο. Επίτροπος πλέον δεν υπάρχει, θα αντικατασταθεί. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν κυρία Κοντά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η τελετή που έλαβε χώρα την προηγούμενη Δευτέρα στο Θέατρο Φλαζέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα παρακολουθήσουμε το θέμα αυτό των βραβείων με μεγάλη προσοχή. Κυρία Κοντά, θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση, αλλά και να δούμε και τις προοπτικές για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας, γιατί πιστεύω ότι η συνεργασία μεταξύ Επιτρόπου, Επιτροπής και της δικής σας Επιτροπής Πολιτισμού του Κοινοβουλίου είναι επικοδομητική και χρήσιμη και ελπίζω να μπορέσουμε να την ενδυναμώσουμε και να την συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι η συνάντηση λαμβάνει χώρα ακριβώς μετά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία, γιατί αν συνεχιστεί η διαδικασία κύρωσης με τρόπο θετικό, με τους φίλους μας τους Τσέχους, βλέπουμε μια ενδυνάμωση κάποιων δράσεων, κάποιων ενεργειών. Πρώτον, όσον αφορά τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον, στον πολύ σημαντικό τομέα των αθλητικών κέντρων, όπου για πρώτη φορά θα υπάρξει κοινοτική αρμοδιότητα. Όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, από τα τρία θέματα που μας απασχολούν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε την εφαρμογή του τριγώνου της γνώσης με τρεις πτυχές εκπαίδευσης. Μετά θα αναφερθώ στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα κύρια θέματα που έχουμε προχωρήσει το 2009 και θα ολοκληρώσω με τις νέες μας πρωτοβουλίες, νέες θεματικές πρωτοβουλίες που θα σας απασχολήσουν φέτος. Ξεκινάω λοιπόν από το τρίγωνο της γνώσης. Θα προσπαθήσω εδώ να αναφερθώ σε τρία θέματα. Το πρώτο νομίζω ότι ήταν ε, πάρα πολύ σημαντικό και ήταν η έγκριση ενός νέου πλαισίου στρατηγικής για την συνεργασία μας σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτό έγινε υπό την Τσεχική Προεδρία. Πολύ ξεκάθαρα δείχνει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση βρίσκονται στο κέντρο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Και άρα έτσι μπορούμε να προετοιμαστούμε για τη συνέχεια, για την περίοδο μετά τη Λισαβόνα, μετά το 2010. Γιατί η στρατηγική που έχει υιοθετηθεί είναι εκπαίδευση και κατάρτιση ενώπιση του 2020. Οι προτεραιότητε είναι εξή. Πρώτον, ποιότητα και αποτελεσματικότητα, η αριστεία δηλαδή που λέμε των πολιτικών παιδείας. Δεύτερη προτεραιότητα είναι η ισότητα και τα δικαιώματα του πολίτη. Είναι ο ρόλος υπέρ της κοινωνικής συνοχής και ο τρίτος τομέας ίσως είναι πιο νέος όσον αφορά τις σκέψεις μας για την πολιτική παιδεία, είναι η καινοτομία και η δημιουργία. Ο ρόλος των συστημάτων εκπαίδευσης βέβαια είναι πολύ σημαντικός για να έχουμε μια πιο καινοτόμα και πιο δημιουργική Ευρώπη. Και όλα αυτά βέβαια μέσα στην προοπτική της διαβίου κατάρτισης υπογραμμίζοντας όλος ιδιαίτερος την κινητικότητα. Και όχι μόνο για τα προγράμματα, στα οποία θα επανέλθω και μετά, αλλά όσον αφορά μια πολιτική κινητικότητα πιο δυνατή από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Και για την απασχολησιμότητα που αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τα συστήματα εκπαίδευσης που έχουμε. Χάρη λοιπόν σε αυτό το νέο πιο φιλόδοξο πλαίσιο, θα έπρεπε να μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα με το πλαίσιο που ολοκληρώνεται το 2010. Ε, τα σημεία αναφοράς μας θα τα προσαρμόσουμε. Έτσι ώστε για πρώτη φορά να έχουμε benchmarks και στον τομέα της κινητικότητας και να δούμε μήπως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παράγοντας απασχολησιμότητας. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε συνεχή διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή αυτού του πλαισίου συνεργασίας. Με τα κράτη-μέλη βέβαια. Αλλά εσείς, οι ιδέες σας η προσέγγισή σας πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το τομέα. Ίσως αυτή είναι η πρώτη μεγάλη πρόοδος που πετύχαμε στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσα στο 2009. Το δεύτερο στοιχείο είναι ο διάλογος μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Άκουγα νωρίτερα στα πλαίσια των μελετών ότι αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο υπάρχει δουλειά να γίνει. Ε, λοιπόν, η Κομισιόν ξεκίνησε ένα μόνιμο φόρουμ διαλόγου ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις. Στρέφεται γύρω από τρία θέματα. Τα κουρίκολομ, η μέθοδοι και ο τρόπος εταιρικής σχέσης, κάτι αρκετά περίπλοκο, και νέες ε, νέα προσόντα που χρειάζονται για τις νέες θέσεις απασχόλησης. Καταλήξαμε σε μια ανακοίνωση η οποία προβλέπει να επεκταθεί η συνεργασία αυτή. Και αυτό είναι κάτι που το ζητάνε επιχειρήσεις. Να επεκταθεί λοιπόν πέρα από τα πανεπιστήμια η συνεργασία, να γίνεται και με τα σχολεία. Και ξέρω το κόμινους είναι δικό σας παιδί λιγάκι κυρία Πρόεδρε το Communist ρέγγιο κυρίως, που αποτελεί βάση για τέτοιου είδους συνεργασία. Θα φροντίσουμε λοιπόν να ενισχυθεί αυτός ο διάλογος. Το τρίτο στοιχείο τώρα, όπου είναι η Επιτροπή Ήτρε κυρίως, που ενδιαφέρθηκε, αλλά και εσείς βέβαια, ιδιαίτερως εσείς κυρία Πρόεδρε, είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Αποτέλεσε αντικείμενο μεγάλων συζητήσεων το 2008 και στις αρχές του 2009. Ή ε, λοιπόν, τώρα το Ευρωπαϊκό Αυτό Ινστιτούτο αρχίζει να λειτουργεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιλέξει το Δεκέμβριο τις πρώτες κοινότητες γνώσης και καινοτομίας που αποτέλεσαν αντικείμενο προτάσεων που είχαν να κάνουν με τις κλιματικές αλλαγές, με τις βιώσιμες ενέργειες και με την τεχνολογία της γνώσης. Ορίστηκε διευθυντής μόλις, που σημαίνει ότι σιγά σιγά γίνεται αυτόνομο το Ινστιτούτο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο τρίγωνο της γνώσης, και παραδοσιακά όταν μιλάμε γι' αυτό, τελειώνουμε με την έρευνα και την καινοτομία. Ε, λοιπόν, η εκπαίδευση, περισσότερο σήμερα από ό,τι κατά το παρελθόν, παίρνει τη θέση που της πρέπει. Και το βλέπουμε αυτό και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Εκεί το Διοικητικό Συμβούλιο επέμεινε πάρα πολύ για το σημαντικό ρόλο που παίζει η εκπαίδευση. Το δεύτερο θέμα, το οποίο ήθελα να αναφέρω, είναι οι εξελίξεις που είχαμε το 2009. Το ξέρετε βέβαια ότι είχαμε το πακέτο επιτροπολογίας. Το πακέτο επιτροπολογίας μας επέτρεψε να ανταποκριθούμε σε μια ανησυχία που είχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ήθελε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τη διαχείριση προγραμμάτων που έχει η διευθυνσή μου. Τα πέντε προγράμματα. Θέλατε επίσης να αποφασίζονται πολύ πιο γρήγορα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρίως για τις μικρές δομές που συμμετέχουν στα προγράμματά μας το εκτελεστικό όργανο που εξαρτιέται από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού και Παιδείας δούλεψε πολύ για να διασφαλιστεί η απλοποίηση. Ορισμένοι από εσά και εσείς κύριε Πρόεδρε πήγατε. Αν η Επιτροπή σας θέλει να επισκεφθεί και πάλι την υπηρεσία αυτή θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα και με τις υποψηφιότητες και με τη διαφάνεια της επιλογής, της διαδικασίας επιλογής. Για το κομμάτι εκπαίδευση. Εδώ έχουμε δύο σημαντικές εξελίξεις το 2009. Το πρώτο ήταν η εξωτερική διάσταση της συνεργασίας. Δηλαδή συνεργαζόμαστε και εκτός Ευρώπης μέσω το Erasmus Mundus 2 σε συναπόφαση μαζί σας. Το στηρίξατε. Από το Φεβρουάριο λοιπόν του 2009 έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μας επιτρέπει να αυξάνουμε την προβολή του σε τρίτες χώρες. Αν δούμε τους δικαιούχους τελικά διαπιστώνουμε ότι έχουμε Ινστιτούτα Αριστείας πολύ περισσότερα από ό,τι κατά το παρελθόν. Ενισχύσαμε και τον πολιτικό διάλογο με ορισμένες χώρες. Κίνα, Ινδία, Ενωμένες Πολιτείες, θα πάω σε δύο μέρες, ε, Βραζιλία, Μεξικό. Η ευρωπαϊκή δηλαδή ανώτατη εκπαίδευση γίνεται πιο ελκυστική προς τα έξω. Έχουμε και την πρώτη εταιρική σχέση Comenius Regio, που είναι δικιά σας πρωτοβουλία κύριε Πρόεδρε. 450 περιφέρειες κατέθεσαν έτοιμα ε, για χρηματοδότηση. Οι περισσότερες από τις μισές θα υιοθετηθούν. Και στο τέλος της ε, χρονιάς θα έχουμε συγκεντρώσει τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις. Και να ξέρετε ότι οι περιφέρειες πολύ ένθερμα υποστήριξαν αυτές τις πρωτοβουλίες. Μην ξεχνάτε και το Erasmus για τους μαθητευόμενους, που ήταν επίσης πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου. στα πλαίσια του προγράμματος Λεωνάρντο. Βοήθησε στην κινητικότητα των μαθητευόμενων, γιατί η κινητικότητά τους αυτή πήρε μεγαλύτερη διάσταση. Τώρα το Ευρωπαϊκό Έτος για την δημιουργία και την ε, καινοτομία. Μεγάλη επιτυχία. Θα ακούσατε τον ε, κύριο Μπαρόζο στο Φόρουμ για τον Πολιτισμό που είπε ότι είναι μια από τις μεγάλες μας επιτυχίες. Βλέπετε υπάρχει, ε, είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο, η καινοτομία και η δημιουργία. Οι επιχειρήσεις και ο πολιτισμός έχουν σχέση μεταξύ τους, γιατί υπάρχει στις επιχειρήσεις καινοτομία και ε, στον πολιτισμό υπάρχουν επιχειρήσεις. Έχουμε πρέσβεις για φέτος, είτε πρόκειται για τι μέρες και και άλλους, όλοι αυτοί τον Νοέμβριο θα δώσουν ένα μανιφέστο που θα λέει τι πιστεύουν ότι πρέπει να περιλαμβάνει η δημιουργία και η καινοτομία. Είναι οι πρέσβεις δημιουργίας μας, όπως τους λέμε, και καινοτομίας. Έτσι πιστεύω ότι θα βάλουμε τις βάσεις για μια πιο μακροπρόθεσμη πολιτική. Έρχομαι τώρα στον πολιτισμό. Το 2009 ήταν μια σημαντική χρονιά. Δεν θα μπω στο θέμα της πολυγλωσσίας. Ο Επίτροπος Ορμπάν θα έρθει αύριο να σας μιλήσει γι' αυτό. Στον πολιτισμό, αυτό κάθε αυτό θα επικεντρωθώ. Αναφερθήκατε στο φόρουμ που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα στην πλατεία Φλαζέ. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, πιστεύω. Πολλοί κόσμος από τον πολιτισμό ήρθε και αναγνώρισε ότι είχε επιτευχθεί σημαντική πρόοδο στα θέματα του πολιτισμού, γιατί μην ξεχνάμε δεν υπήρχε πολιτισμική πολιτική. Τώρα υπάρχει ατζέντα για τον πολιτισμό. Αλλά βέβαια πολλά μένει να γίνουν ώστε να βρεθεί στο κέντρο ο πολιτισμός. Και κυρίως στο κέντρο της οικονομικής πολιτικής. Υπάρχει και το βραβείο για τη λογοτεχνία το ευρωπαϊκό. Και αυτό είναι σημαντικό για να δώσουμε μεγαλύτερη προβολή στον πολιτισμό. Τα νέα ταλέντα που κέρδισαν αναγνωρίστηκαν ότι είναι μεγάλης ποιότητας. Θα έχουμε τώρα και δύο πρωτοβουλίες, ναι, στον τομέα αυτό του πολιτισμού, που και δύο έχουν να κάνουν με δύο σημαντικές πτυχές του πολιτισμού. Είναι ο πολιτισμός ως κινητήριος δύναμης της διαφοροποίησης αλλά και της ενότητας της Ευρώπης, η ψυχή της Ευρώπης, Και από αυτού, αρχές της επόμενης χρονιάς θα έχουμε πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το λεγόμενο σήμα της Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς. Είναι κάτι που υποστήριξε το Κοινοβούλιο ήδη από το 2007. Τώρα θα γίνει ευρωπαϊκό σήμα, μια ευρωπαϊκή δράση. Κάτι σαν τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πολιτισμού και θα είναι πιστεύω κάτι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες την ε, ευρωπαϊκή κληρονομιά. Το άλλο είναι κινητήρια δύναμη για την οικονομία, ο πολιτισμός. Κάναμε μελέτη που δείχνει ότι 10% του ΕΠ έχει να κάνει με την δημιουργία και τον πολιτισμό. Υπάρχει πράσινη βίβλος λοιπόν για τις δυνατότητες που έχει ο πολιτισμός και του χρόνου θα κάνουμε συγκεκριμένη πρόταση όπου ακριβώς συνδέουμε τον πολιτισμό με τις επιχειρήσεις μέσω της στρατηγικής ανάπτυξης και απασχόλησης. Και για να επανέλθω λίγο στο μήνυμα που έδωσε ο Βιν Βέντερς στο τέλος του φόρουμ, που είπε ότι ο πολιτισμός είναι η κινητήρια δύναμη της Υπήρου. Ε, νομίζω ότι αυτό συλλογικά σε όλα τα κοινοτικά όργανα δίνει ό,τι στοιχεία χρειαζόμαστε για να αναπτύξουμε περισσότερο την πτυχή πολιτισμός. Άρα λοιπόν 2010 και μετά πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το ευρωπαϊκό σήμα κληρονομιάς και πάνω στις δημιουργικές επιχειρήσεις. Τώρα μια που είμαστε και στην πολυγλωσία θα περάσω στα αγγλικά. Έχουμε πολλές κοινέ προκλήσεις για το μέλλον. Η πρώτη έχει να κάνει με την ε, χρήση. Το 2009 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η νεότητα. Πώς ε, οι νέοι θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος. Την απασχόληση βέβαια, πρώτα απ' όλα, που είναι πολύ βασικό. Αλλά επίσης θέλουμε την δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα, την ε, κοινωνική συμμετοχή, τη συμμετοχή των πολιτών ε, και τον εθελοντισμό για τους νέους. Αυτές είναι προτάσεις που προχωράνε σε όλα τα φόρα των νέων. Έχουμε κάνει διαβουλεύσεις με τους νέους και ήδη το Φεβρουάριο του 2009 είχαμε εδώ τους νέους, οι οποίοι συνεισέφεραν πολύ σημαντικά στην εκπόνηση της στρατηγικής μας. Σήμερα πια περιμένουμε τις απόψεις σας και του Συμβουλίου που πρέπει να υιοθετήσει τη στρατηγική αυτή στην επόμενη συνεδρίασή του τον Νοέμβριο. Νομίζω ότι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για τη στρατηγική αυτή είναι ο διάλογος με τους νέους. Είμαστε στη διαδικασία να αποφασίσουμε για την νέα πρωτοβουλία μέσα σε νέα πλαίσια διαλόγου με τους νέους. Είναι όλο και πιο σημαντικό αυτό μέσα στην οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε και στις δυσκολίες που έχουν οι νέοι να να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Βασιζόμαστε σε καλή συνεργασία μαζί σας, γιατί εσείς ήσασταν στοιχείο κλειδί το 2008, όταν οργανώσαμε εκείνη την εβδομάδα που συναντηθήκαμε με τους νέους. Θα είμαστε συνέχεια σε επαφή μαζί σας για να οργανώσουμε την επόμενη τέτοια εβδομάδα νέων. Δεύτερο θέμα, κινητικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει πράσινη βίβλο για την κινητικότητα των νέων. Βασίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπογαλλικής Προεδρίας το 2008. Εκεί έλεγαν ότι η κινητικότητα πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση και ότι ο κάθε νέος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πάει στο εξωτερικό. Αργότερα, εντάξει υπάρχει και το έρασμος βέβαια που είναι το πιο γνωστό μέσο που διαθέτουμε, αλλά αυτό να ισχύει και σε εθελοντική βάση, με ανταλλαγές μεταξύ νέων. Οπότε, έχουμε ξεκινήσει με αυτή την πράσινη βίβλο γιατί θέλουμε να δούμε πώς θα αυξήσουμε τις δυνατότητες που έχουν οι νέοι για κινητικότητα. Να αποτελέσει τον κανόνα δηλαδή κινητικότητα. Και η ανταγωνιστικότητα βέβαια μας ενδιαφέρει, που αποτελεί πτυχή της κινητικότητας και θέλουμε όλους τους νέους μαθητευόμενους, Φοιτητέ. όλους τους νέους να δούμε πώς θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να πάνε στο εξωτερικό. Δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2009 η πράσινη αυτή βίβλος. Μας βοήθησαν πολλοί εταίροι και θα δείτε ότι συμπεριλαμβάνεται και στις κατευθυντήριες γραμμές του Πρόεδρου Μπαρόσο, όπου προτείνει την πρωτοβουλία που την ονομάζει η νεότητα εν κινήσει. Είναι μια πρωτοβουλία πολιτικής για να πάμε πιο κοντά στην κινητικότητα των νέων, να την ενισχύσουμε και τα Υπουργεία στα πλαίσια της Μπολόνια συμφώνησαν με το στόχο του 20% το 2020 κινητικότητα για τους νέους. Το τελευταίο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι κάτι για το οποίο το Κοινοβούλιο πιέζει εδώ και πολύ καιρό. Έχει να κάνει με τον εθελοντισμό. Τον Ιούνιο του 2011 προτείνουμε να είναι Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Για πρώτη φορά βλέπουμε τον εθελοντισμό σαν κάτι το οποίο έχει να κάνει με όλες τις πτυχές της πολιτικής μας και αφορά όλα τα στρώματα της κοινωνίας, όχι μόνο τους νέους, όχι μόνο τους ηλικιωμένους, αλλά ολόκληρο τον πληθυσμό. Η πρόταση βασίζεται σε ανάλυση που έγινε και που δείχνει ότι ο εθελοντισμός αποτελεί κάτι πολύ σημαντικό για το μέλλον και εσείς τον Μάρτιο του 2008 υιοθετήσατε σχετική έκθεση και λέτε ότι ο εθελοντισμός συνεισφέρει στην οικονομική και την κοινωνική συνοχή. Ε, περιοριστήκαμε στο άρθρο 308 της συνθήκης ως νομική βάση, αναγκαστήκαμε. Αλλά βέβαια το κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό για μας και γι' αυτό έχουμε προβλέψει ένα ειδικό άρθρο, το άρθρο 5, για την... ώστε να υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας όταν πρόκειται για την απόφαση. Και χαίρομαι που και το Συμβούλιο ε, δείχνει να δέχεται μια πολιτική συμφωνία πάνω στην πρόταση αυτή και να την υιοθετήσει τον Νοέμβριο. Ελπίζω ότι και το Κοινοβούλιο θα στηρίξει την πρόταση για το ευρωπαϊκό αυτό έτος. Γιατί άμα το θέλουμε όντως το 2011 πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσω. Η διαδικασία είναι μακρά. Εν κατακλείδη λοιπόν. Θέλω να υπογραμμίσω ότι όχι μόνο το 2009 ήταν ζωτική σημασία για την Ευρώπη, είχαμε και τις ευρωεκλογέ και ξέρουμε τι γίνεται και με την Επιτροπή, τα δημοψηφίσματα. Από την άλλη μεριά όμως ήταν και μια χρονιά πολύ θετική όσον αφορά τα θέματα της Επιτροπής σας. Το 2010 είναι πολλά υποσχόμενο. Θα αποτελέσει πρόκληση για τους πολίτες όσον αφορά την απασχόληση και την ανάπτυξη. Είναι ζωτική σημασία λοιπόν να συνεργαστούμε για να πετύχουμε πρόοδο και στην ανταγωνιστικότητα και στην εκπαίδευση, αλλά και όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών και τον ενθουσιασμό τους απέναντι στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν κυρία Πρόεδρε και είμαι στη διαθεσή σας για ό,τι ερωτήσεις, κριτική ή σχόλια έχετε. Ευχαριστώ κυρία Κοντά. Πολύ συνοπτικά, πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε. Πρώτα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους οι οποίοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Ο κύριος Φίζας Οξέλα. Eh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τη Γενική Διευθύντρια που ήρθε εδώ και μας έδωσε τόσες εξηγήσεις. Τα θέματα πολιτισμού με ενδιαφέρουν όλους ιδιαίτερους και έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Όσον αφορά αυτό το σήμα, το ευρωπαϊκό, στο οποίο αναφέρθηκε, πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρουσα ιδέα αλλά πρέπει να δούμε τι διαφορά μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στο σήμα αυτό και τα σήματα που δίνει η UNESCO που ορίζει ως πολιτιστική κληρονομιά κάποια έργα. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι διαφορά θα υπάρχει. Επίσης θέλω να αναφερθώ και στην επικοινωνία. Θα έπρεπε να υπάρξει μια εκστρατεία ενημέρωσης για να ξέρουμε ποια είναι αυτά τα σημεία που παίρνουν αυτό το ευρωπαϊκό σήμα. Είναι πολύ σημαντικό κάτι τέτοιο και για τον τουρισμό μας και για την οικονομική ε, πρόθεση. Πώς δίνονται τα σήματα αυτά, πώς θα δίνονται τα σήματα ευρωπαϊκής κληρονομιάς μετά από πρόταση των κρατών μελών, ε, περνάει κάθε πρόταση από κάποια φίλτρα της Κομισιόν του Κοινοβουλίου, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Και ω συνέχεια τη πρώτη μου ερώτηση να πω ότι πιστεύω πως ο ευρωπαϊκός πολιτισμός πρέπει να αποτελεί πρέσβη σε ολόκληρο τον κόσμο που να προωθεί την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ήπειρος που μπορεί να πει ότι περισσότερο από εμά πολιτιστικά στοιχεία, ε, μνημεία κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν πολύ καλό να δούμε και το άλλο. Όταν μιλήσαμε για την μαθητεία και για το Εράσμους, μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και για τους νέους δημιουργούς που να μπορούν να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό που έχουμε δηλαδή για τους φοιτητές να το κάνουμε και για τη δημιουργία. Έτσι οι νέοι μπορούν να πλουτίσουν τις εμπειρίες τους σε άλλα πολιτισμικά πλαίσια, σε άλλες χώρες. Αναφερθήκαμε και για την κινητικότητα των νέων. Να προσθέσουμε και των δημιουργών. Γιατί υπάρχουν νέοι που συμμετέχουν σε μια ορχήστρα, για παράδειγμα. Εντάξει, πάνε από μια χώρα στην άλλη, μιλάνε με τους ομολόγους τους. Υπάρχουν όμως προβλήματα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτά πώς λύνονται τα ζητήματα. Πάντως όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, ιδίω τώρα που προβλέπεται η έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας, μπορούμε να προχωρήσουμε και στο θέμα του αθλητισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Σκαβαντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά όταν ακούει κανείς την κυρία Κοντά να μιλάει για τις προοπτικές των επόμενων μηνών, να κάνει έναν απολογισμό χαίρεται ιδιαίτερα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να επαναλάβουμε άλλη μια φορά ότι πραγματικά ο πολιτισμός θα πρέπει να προϋπάρχει κάποιων πολιτικών και οικονομικών διαπραγματεύσεων. Εν πάση περιπτώσει, ο προϋπολογισμός δεν μας βοηθάει. Αλλά αν κοιτάξει κανείς τη συνδίκη της Λισαβόνας, βλέπει ότι υπάρχουν κάποιες δυνατότητες. Κυρία Κοντά, θα πρέπει να μας στηρίξετε, να δείξουμε και κάποια φαντασία. Εμείς θα ασκήσουμε πίεση πολιτική, έτσι ώστε να προχωρήσουν αυτές οι δυνατότητες. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι διαπιστώνουμε πάντα όταν ο πολιτισμός λείπει από ένα πολιτικό πρόγραμμα, διαπιστώνουμε πόσο ε, ομές και στεγνές είναι οι πολιτικές. Ήμουν στην ε, Ιρλανδία και έμεινα τρεις μέρες για το δημοψήφισμα και συνειδητοποίησα πόσο σημαντική είναι η ιδιαιτερότητα της κάθε χώρας ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ιρλανδίας. Κάτι που πραγματικά μας βοηθάει όλους και μας που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η Ιρλανδία μας προσφέρει κάτι, μια πρωτοτυπία στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Και θα ήθελα εδώ να πω, κυρία Πρόεδρε, ότι εκ παραλίλου με τη συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε αυτού του είδους τις ακροάσεις, σαν και αυτή που οργανώσατε το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο αυτού του χρόνου. Γιατί δεν ακούγονται αρκετά οι καλλιτέχνες. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που έγινε στο φόρουμ, αλλά πιστεύω ότι και εδώ που λαμβάνονται οι αποφάσεις θα πρέπει οι καλλιτέχνε, οι δημιουργοί, αλλά και οι ερευνητές να αποκτήσουν μια πιο ισχυρή θέση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φεράιν. Καταρχήν, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πάρα πολύ σημαντική σας παρουσίαση. Μιλήσατε για τους νέους, για την επαγγελματική κατάρτιση των νέων. Και αυτό είναι κάτι που ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές αντιμετωπίζουν οι νέοι, οι φοιτητές, οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα. Επειδή όμως υπάρχουν τελείως διαφορετικά συστήματα κατάρτισης, ε, συνεχίζουν να υπάρχουν εμπόδια για τους νέους αυτούς οι οποίοι θέλουν να κινηθούν στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ θετικό αυτό που μας λέτε, ότι στο μέλλον αυτά τα εμπόδια θα εξαλειφθούν και ότι θα μπορέσει να υπάρξει αυτή η γέφυρα μεταξύ του συστήματος του εκπαιδευτικού και του βιομηχανικού τομέα, του κόσμου της οικονομίας και αυτό ιδιαίτερα για τους νέους που έχουν διαφορετικά πρότυπα και εκπαιδευτικά αλλά και κατάρτισης επαγγελματικής. Η Πρόεδρος, και εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Μιλήσατε για τη συνεργασία μεταξύ του κόσμου των επιχειρήσεων και των πανεπιστημίων. Μιλήσαμε επίσης για το θέμα των εκπαιδευτικών συστημάτων. Είναι θέμα επικουρικότητας. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε εδώ χωρίς να κάνουμε αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε, λέει η Πρόεδρος. Δεύτερη ερώτηση. Κομμένιου Ρέγγιο. Μπορείτε να μας δώσετε ένα ή δύο παραδείγματα πώς αυτό το πρόγραμμα Ρέγγιο λειτουργεί. Είπατε ότι είχε πολύ καλή αποδοχή. Τρίτη ερώτηση. Πάρα πολλά πράγματα εμπόδισαν τις προτάσεις της Επιτροπής να προχωρήσουν σε θέματα κατάρτισης. Πολλά όμως προχώρησαν χωρίς να υπάρχουν οι πραγματικές αρμοδιότητες. Έχω πολλά παραδείγματα. Και η ερώτησή μου είναι το θέμα της διδασκαλίας, το θέμα των καθηγητών, των δασκάλων, μπορείτε να το πλαισιώσετε έτσι ώστε να αποκτήσει πάρα πολύ σοβαρή, αν θέλετε, θέση, όχι υποθάλποντας την έρευνα. Και η έρευνα και οι ερευνητέ είναι πάρα πολύ σημαντικοί, αλλά οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και η διδασκαλία. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε και αυτό το τομέα. Έκανα τρεις ερωτήσεις. Κυρία Κοντά, ας απαντήσουμε πρώτα και κατόπιν ε, θα δώσω το λόγο και στους υπόλοιπους συναδέλφους για να απαντήσουν. Για να κάνουν τις ερωτήσεις, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν, ε, ας αναφερθώ στις ερωτήσεις και στα σχόλια. Κύριε Ξέλα, και καταρχήν η χώρα σας, η Ισπανία, είναι, ε, ζητά ιδιαίτερα έντονα να μπορέσουμε να έχουμε αυτήν την αυτό το σήμα υπό την ε, Ισπανική ε, Προεδρία είναι η είναι η χώρα η Ισπανία που ξεκίνησε αυτό το ε, σήμα, όπως έχει τώρα, δηλαδή σε διακυβερνητικό επίπεδο. Προστιθέμενη αξία σε σχέση με το σήμα της UNESCO αποτέλεσε αντικείμενο ατερμόνων συζητήσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το βασικό κριτήριο σε αυτό το πλαίσιο και θα δούμε ποια θα είναι η επίσημη πρόταση της Κομισιόν και οι αποφάσεις που εσείς και το Συμβούλιο θα λάβετε, πάντως ε, είναι να συνδέεται άμεσα με την ευρωπαϊκή ιστορία και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Και να δώσω δύο πολύ διαφορετικά παραδείγματα δύο χωρών που στο πλαίσιο αυτό του διακυβερνητικού σήματος έχουν εντοπίσει σήματα που είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που, τύπου της UNESCO είναι η Πολωνία με το ναυπηγείο του Γκτάνσκ και η Γαλλία με το UNI. Είναι δύο διαφορετικές ιστορικές περίοδοι που συνδυάζονται με το προσκύνημα και το ε, ε, οναστικές τάξεις για τη Γαλλία και για την ε, Πολωνία με την παράδοση. Ε, αυτά λοιπόν μπορεί να δώσουν μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αξι, προστιθέμενη αξία. Εσεί και το Συμβούλιο θα αποφασίσετε βέβαια από αυτόν όταν ε, με τη βάση της πρόταση τη Κομισιόν θα ολοκληρώσετε την προσέγγιση. Και περιμένω περίπλοκου ε, ορισμού, γιατί υπάρχουν διαφορετικέ απόψει για το ρόλο που μπορεί να παίξει κάθε χώρα στο πλαίσιο αυτό. Για το έρασμο των μαθητευομένων και, των νέων δημιουργών. Το έρασμο είναι επίση ένα σήμα πολύ καρποφόρο έρασμο για πολλούς πολύ κόσμο έχει αποφέρει καρπούς. Ας πούμε, ε, για τους επιχειρηματίες έγινε έρασμος, για τους στατιωτικούς έγινε έρασμος. Ε, είναι η αρχή της κινητικότητας βασικά. Νομίζω πως όντως οι νέοι δημιουργοί είναι μια πολύ σημαντική ομάδα στο πλαίσιο αυτό. Και οι πιλωτικές δράσεις που υιοθέτησε το προηγούμενο κοινοβούλιο θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε για τους καλλιτέχνες γενικότερα τις δυνατότητες κινητικότητας, γνωρίζοντας τα εμπόδια, τα γνωρίζουμε όλα τα εμπόδια στην κινητικότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και είναι πιο περίπλοκο όταν έχουμε καθεστώς ανεξάρτητο επαγγελματία. Είναι κάτι δηλαδή που οι πιλωτικές αυτές δράσεις θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε και σε αυτό το επίπεδο της ανάλυσης. Τώρα, για τα σχόλια του κ. Καβαντά. Πιστεύω πως ο πρόεδρος Μπαρόζο τόπε τη στιγμή της απονομής του βραβείου λογοτεχνίας, ότι ο πολιτισμός ξεπερνά την οικονομία. Αν και η οικονομία είναι θεμελιώδης και όλες οι προκλήσεις ε, που έχουμε και η μεγάλη συζήτηση είναι εδώ είναι αυτό που λέμε σε ωραία γαλλικά το mainstreaming της κουλτούρας, δηλαδή το να λαμβάνεται υπόψη ο πολιτισμός σε όλες τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών πολιτικών της Ένωσης. Και επίσης αληθεύει ότι ο πολιτισμός ενθουσιάζει τον κόσμο πολύ περισσότερο από ότι η εσωτερική αγορά ή οι κανόνες του ανταγωνισμού. Όσο και αν είναι σημαντική όλη αυτή. Κινητοποίηση λοιπόν των πολιτών είναι ένας από τους στόχους του φόρουμ. Ωστόσο, και νομίζω πως εν, λό, εν μέρη αυτό επετεύχθη, δεν βλέπουμε αρκετά τους καλλιτέχνες τους ίδιους. Ο κόσμος, η κοινωνία των πολιτών, οι διάφορες πολιτιστικές δομές, κάποιοι καλλιτέχνες. Ο Βιμβέντρες είναι ένα παράδειγμα. Είχαμε τον ε, και διάφορους άλλους στο φόρουμ πάντως, το να ακούσουμε τη φωνή των καλλιτεχνών είναι ένας από τα σημαντικές προκλήσεις για το μέλλον. Και φυσικά η πολιτιστική διαφοροποίηση που αντιπροσωπεύει η Ιρλανδική περίπτωση. Ε, είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλη, μεγάλη πρόκληση ευρωπαϊκή γιατί η Ευρώπη έφερε, πρόθεσε την σύμβαση της UNESCO για την πολιτιστική πολυμορφία τόσο εντό όσο και εκτός. Ευρώπης. Η συμφωνία Καρικόμ που κάναμε με διάφορους εταίρους ε, από τις χώρες της Καραϊβικής και του Ειρηνικού είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Αυτά λοιπόν αγγίζουν την καρδιά της Ευρώπης. Ναι, προεπαγγελματική δραστηριότητα και εδώ διαπιστώνουμε έχουν πολύ δύσκολο βέβαια να έχουμε στοιχεία για την κινητικότητα, για την κατάρτιση, αλλά σίγουρα είναι λιγότεροι από ό,τι για τα πανεπιστήμια. Και υπάρχουν και κάποια ευρωπαϊκά μέσα, soft law, που υιοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια, υπάρχει το πλαίσιο της αντιστοιχίας των πτυχίων, επιτρέπει δηλαδή τη διαφάνεια ιδιαίτερα όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και δύο ακόμα μέσα, το ΕΚΒΕΤ, δηλαδή η πίστοση μεταφορά στο τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και το ΕΚΑΦ, δηλαδή ασφάλεια για την ποιότητα σε θέματα επαγγελματική κατάρτιση, που είναι δύο εργαλεία που επιτρέπουν να διασφαλιστεί η αξιοπιστία τη κατάρτιση πολύ σημαντικό αυτό σε σχέση με τις νέες θέσεις απασχόλησης και ταυτόχρονα διασφαλίζεται η μετάβαση, η μεταφορά μάλλον των πιστώσεων που Ε, αποκτήθηκαν με τη νέα κατάρτιση. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για την κατάρτιση και για την κατάρτιση των ενηλίκων, ε, ειδικά λόγω της εξέλιξης της αγοράς εργασίας, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Για το ερώτημά σας, για την επικουρικότητα, κυρία Πρόεδρε, επικουρικότης. Φυσικά, όταν μιλάμε για βιογραφικό σημείο, δεν είναι η Ένωση, όχι, είναι οι επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια που συζητούν μαζί για τα βιογραφικά. για την ύλη ε, των πανεπιστήμιων. Είναι δύο κόσμοι οι οποίοι καταρχήν δεν συμπαθιούνται μεταξύ τους, αλλά πρέπει όλα ένα και περισσότερο να συνεργάζονται. Πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος, όταν μιλάμε για το τρίγωνο της γνώσης, να ξεχάσουμε την παιδεία. Είναι ένας κίνδυνος που μάλιστα βλέπω να προκύπτει και στις συζητήσεις ε, μέσα στο πλαίσιο της ε, Κομισιόν. Μιλάμε για το τρίγωνο της γνώσης και καταλήγουμε στην έρευνα ε, και την ανάπτυξη. Η έρευνα χωρίς καλό επίπεδο παιδείας και η καινοτομία δεν γίνεται να υπάρξουν. Η παιδεία λοιπόν θα πρέπει να τονιστεί περισσότερο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό κάναμε με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Πιστεύω πως αν οι κοινότητες καινοτομία και της γνώσης αντικατοπτρίζουν ε, καλύτερα αυτό το τρίγωνο και ήταν και ένα σημείο κλειδί των ε, προκηρύξεων που έγιναν από την, ε, από την Κομισιόν, εκεί θα έχουμε ένα εργαλείο σωστό. Και μάλιστα στην τελευταία άτυπη σύνοδο του Συμβουλίου που έγινε πριν από λίγες μέρες στη Στοκχόλμη, έγινε λόγος για το ρόλο κλειδί των ε, διδασκόντων και την κινητικότητα των ε, δασκάλων για να υπάρξει άνοιγμα του διδακτικού προσωπικού και αυτό θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για το Κομένιους, το έρασμος, το Λεωνάρτο που έχουν συνιστώσεις κινητικότητας μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών για την κινητικότητα των διδασκόντων και των ε, υπευθύνων για την κατάρτιση. Θα υπάρξουν αλλαγές πολύ συγκεκριμένες για κάποιες γενναίες των ε, διδασκάλων και γι' αυτό θα πρέπει πιθανότατα να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο σχετικά αφορά την κινητικότητα. Και αυτό περιλαμβάνεται σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτέ οι σκέψει είναι κάπω πρόημος, αλλά είναι χρήσιμο και για τι νέε δημοσιονομικέ προοπτικέ και το πρόγραμμα. Μήπω η κινητικότητα των διδασκάλων θα πρέπει να μπει μέσα στο επίκεντρο των προγραμμάτων. Είναι, ήταν μάλιστα και το μήνυμα του Ισάτυπη Συνόδου της Σουηδίας. Κομμένης λέει η πρόεδρος. Α, συγγνώμη. Ναι, πολιτική γκάφα μόλις έκανα. Είναι πολύ νωρί να το κρίνουμε, γιατί είμαστε ακόμα στο στάδιο τη επιλογής. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι η κινητοποίηση. Αυτή είναι μια θετική πτυχή ότι δηλαδή μόλις είναι λίγο πιο περίπλοκα, όπως είναι το Comenius Regio, ε, κινητοποίησε περισσότερο από 450 δομές και διαφορετικού τύπου εταίρους. Για μένα λοιπόν είναι ήδη ένα, ένα στοιχείο σημαντικό. Θα δούμε τώρα την επιλογή και την ποιότητα των προτάσεων. Πάντως, παρά τον περίπλοκο χαρακτήρα η κινητοποίηση ήταν πολύ έντονη και ήταν έντονη με διαφορετικές δομές. Αν, όπως πιστεύουμε, μπορούμε να επιλέξουμε περίπου το μισό των προτάσεων, πιστεύω πως με 200 προγράμματα θα έχουμε αρκετή μαγιά για να κάνουμε μια πρώτη αξιολόγηση. Τα περισσότερα από τα κράτη-μέλη απάντησαν θετικά στην εκκίνηση του προγράμματος για την ανάπτυξη του Κομένιους 2 για την ε, ατομική κινητικότητα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κέντα. Τρεις ακόμα βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Περνάρα Τράτο και ο κύριος Τσβέρ. Η κυρία Κώστα και η κυρία Νεβεντάλοβα. Εντάξει, θέλει και κάποιος ακόμα το λόγο. Merci, euh, Madame le Commissaire. Ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Η ερώτησή μου είναι... Βεβαίως και Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει ο πολιτισμός να είναι στο κέντρο της συζήτησης και χαίρομαι ιδιαίτερα που σας άξω να το υπογραμμίζετε. Η ερώτησή μου είναι πώς ο πολιτισμός, μάλλον πώς ο, η πολιτική, η πολιτιστική στην Ευρώπη, που θέτει στο κέντρο της τον πολιτισμό, δεν θα θεωρηθεί σαν μια νέα απεικιοκρατία του Βορρά προς τον Νότο. Πώς αντιλαμβάνεται κανείς την ιστορία. Ξέρετε ότι η ιστορία της Ευρώπης είναι συνδεδεμένη με την Αφρική, με τη Βόρεια Αφρική συγκεκριμένα, με το Μαγκρέμπ. Και πώς ενσωματώνεται αυτή τη διάσταση στην πολιτική σας. Πώς η προφορική πολιτιστική παράδοση που δεν διαδίδονται τόσο εύκολα όπως η γραπτή πολιτιστική παράδοση μπορούν να ενσωματωθούν στη σημερινή εποχή. Βγάζω τα γαλλικά εγώ. Hvala za besedo in priložnost, gospa predsednica, da spregovorim in tudi, da se tudi zahvalim gospe Quinten. Da Da se je vela να ευχαριστήσω την κυρία Κοντά για την εξαιρετική της παρουσίαση και τις απαντήσεις που έδωσε μέχρι τώρα στα ερωτήματα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και όλη την ομάδα των συνεργατών της που έχει υποβάλει τόσο εμπεριστατωμένες ε, προτάσεις. Κάποιες πολιτικές που θεωρούνται soft, όπως ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, έχουν πραγματικά λάβει μεγαλύτερη θέση και έχουν ενισχυθεί στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής. Όλοι ξέρουμε όμως ότι συνεχίζουν να υπάρχουν διαφορές, διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, καθώς και μηχανισμοί που τείνουν να ε, να αρμονίσουν λίγο την κατάσταση, όπως παραδείγματος χάρη το σύστημα των πόντων, credits, έτσι ώστε τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και συστήματα κατάρτισης να πλησιάσουν ε, τα ΜΕΝΤΑΔΕ. δε. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά χρειάζεται να υπάρξουν γέφυρες και δυνατότητες περάσματος και συνεργασίας. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε τον κοινό πυρήνα, χωρίς όμως να εξαλείψουμε την πολυμορφία. Κοινέ αξίες ναι, κοινέ αρμοδιότητες, αρμοδιότητες που πρέπει όλοι να διαθέτουν, αλλά χωρίς να εξαλείψουμε, επαναλαμβάνω, την πολυμορφία, αν θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε έναν οικονομικό χώρο που να λειτουργεί. Διαρκώς μιλάμε για τη σημασία της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Θα ήθελα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δείξει πιο απτά αποτελέσματα όταν παραδείγματος χάρη λαμβάνονται οι αποφάσεις για τον προϋπολογισμό. Φέτος τα πράγματα δεν είναι ικανοποιητικά. Ευχαριστώ πολύ. Sì, grazie Presidente. Mi unisco anch'io ai complimenti al direttore per la... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που γίνεται μεγάλη προσπάθεια να τοποθετηθεί ο πολιτισμός στο επίκεντρο των δράσεων, όχι μόνο εδώ στο Κοινοβούλιο ή στην Επιτροπή μας, αλλά σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Έχω μια ερώτηση προς την κυρία Διευθύντρια, μήπως μπορούσε να εμβαθύνει δεδομένης της ε, σημασίας που έδωσε και στο οποίο συμφωνώ στο θέμα της κινητικότητας, αν μπορεί να εμβαθύνει στην έννοια του έρασμος. αν πραγματικά μπορούν να γίνουν επενδύσει σε ορισμένου τομεί, όπω αυτούς που αναφέρθηκαν, όπως ας πούμε το έρασμος για του μαθητευόμενους και όχι ε, ε, ώστε να υπάρξουν πραγματικά ευκαιρίες σε πράγματα, σε θέματα και προγράμματα που μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες. Να μπορέσει έτσι να διεισδύσει μια αντίληψη για μια σημαντική ε, κουλτούρα σε ολόκληρη την Ευρώπη και επίσης επειδή σε επίπεδο των νέων βλέπουμε πως αποτέλεσε αυτό το καλύτερο μέσο για να δημιουργηθούν σχέσεις ανάμεσα στους νέους των διαφόρων εθνών της Ευρώπης. Mrs. Thank you Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και κάτι με ξάφνιασε. Μιλήσατε για τους νέους οι οποίοι θα ήθελαν να βρούνε μια δουλειά ή να περάσουν από κάποια σεμινάρια κατάρτιση στο εξωτερικό η κινητικότητα στους νέους είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο περίπλοκο. Δεν είμαι πεπισμένη ότι αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή να φύγει κάποιο στο εξωτερικό, να έχει ένα πτυχίο από ένα πανεπιστήμιο στη Σλοβακία, παραδείγματος χάρη στη Σλοβακία και να μπορέσει να πάει και να εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μου φαίνεται ότι κάπως αλλιώς θα πρέπει να ιεραρχήσουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Chciałem zapytać, jeżeli można, e, o fragment dotyczący kultury słowa. Mieliśmy okazję, pewnie większość z nas, e, spotkać... Ευχαριστώ. Μιλάμε και για τον παγκόσμιο πολιτισμό, τον πολιτικό του κόσμου. Εμείς συναντηθήκαμε με ομοσπονδίες οι οποίες βρίσκουν απειλή σε αυτό που κάνει το Google ε, με τα βιβλία, τα περιοδικά είναι ένα πολυπλευρές πρόβλημα και περίπλοκο σίγουρο. Από τη μια πρόκειται για τα βιβλία, από την άλλη όμως πρόκειται για τη διάδοση του πολιτισμού, πώς έχουν πρόσβαση δηλαδή όλοι οι πολίτες. Εσείς εκπονείτε καμιά μελέτη, να δείτε με τους εκδότες, με τους ε, καλλιτέχνες, με αυτούς που εκδίδουν περιοδικά επίσης, ποια είναι η γνώμη τους. Εμείς ξέρουμε ότι οι εκδόσεις αυτές χρηματοδοτούνται και η χρηματοδότηση αυτή εξαρτάται από πού προέρχεται, γιατί και αυτό μπορεί να αποκαλέσει απειλή. Αυτό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Και για να τελειώσουμε, η κυρία Κοντά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα απαντήσω σε όλα όσα μου ζητήθηκε. Καταρχήν στην πρώτη ομιλήτρια, όχι δεν πρόκειται για ένα νέο απεικιοκρατικό σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Ατζέντα βασίζεται στον διαπολιτιστικό διάλογο. Φέτος γιορτάζουμε την καινοτομία, τη δημιουργικότητα. Πέρσι όμως γιορτάζαμε τον διαπολιτιστικό διάλογο που ξεκίνησε μάλιστα στη Σλοβενία. Ήσασταν τότε υπουργό Πολιτισμού και νομίζω ήσασταν παρόν. Ο διαπολιτιστικός διάλογος δεν είναι εύκολος σε όλες τις χώρες και αυτό είναι αν θέλετε το θεμέλιο αυτής της ε, ιδέας. Ανοχή, ανταλλαγή απόψεων και πραγματικός διάλογος. Ένας από τους κύριους στόχους αυτής της πολιτιστικής ατζέντα που αποφασίστηκε το 2007 είναι η πρόθεση της πολυμορφίας στον πολιτισμό. Και πολλά από τα σχέδια και τα προγράμματα που στηρίζουμε στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προγράμματα που έχουν σαν θέμα αυτό το πολιτιστικό διάλογο με νέους δημιουργούς. Μάλιστα πολλοί από αυτούς που προέρχονται από τους μετανάστες Ευρωπαίους, έτσι ώστε να γίνει σεβαστή η ισότητα και η ίση πρόσβαση στον πολιτισμό. Όσον αφορά τη Βόρεια Αφρική, στα πλαίσια της Μεσογειακής Ένωσης και της διαδικασίας της Βαρκελόνης, υπάρχει ένα νέο κεφάλαιο για την συνεργασία την πολιτιστική. Την επεξεργαζόμαστε εξάλλου, αυτή την πολιτική, ακόμα. Υπάρχει όμως και η Ανατολική Ευρώπη. Και εκεί χρειάζεται συνεργασία. Και εδώ υπάρχουν ε, κάποιες ιδιαιτερότητες όσον αφορά την εταιρική σχέση προς Ανατολάς, στις γειτονικέ χώρες και 30 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί ήδη σε πολιτιστικά προγράμματα για τις χώρες ΑΚΕ. Ένα μεγάλο φόρουμ που οργάνωσε η Γενική Διεύθυνση η δική μου και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης συγκέντρωσε φορείς ενεργού στον τομέα του πολιτισμού για να ξεκινήσει αυτή η συνεργασία. Αναφέρθηκα προηγουμένω στη συνεργασία Κάριτουμ που είναι, αν θέλετε, η πρώτη απτή ε, απόδειξη ότι αυτή η συνεργασία στον πολιτισμό λειτουργεί. Αυτό συνεχίστηκε εξάλλου στο πρόσφατο φόρουμ. Ο κύριος Σβέα είπε ότι υπάρχουν αυτές οι soft πολιτικές. Έχετε δίκιο. Είναι, αν θέλετε, τομείς της επικουρικότητας, όπως ε, η παιδεία. Η λεγόμενη soft νομοθεσία, όσον αφορά ΕΚΒΕΤ, ΕΚΑΡ, την πιστοποίηση. Όλες αυτές οι ενέργειες στηρίζουν την αμοιβαία αναγνώριση και τη σύγκληση με εκπαιδευτικά συστήματα που είναι μεν διαφορετικά αλλά αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν της ευρωπαϊκής συνεργασίας μας επέτρεψαν να προχωρήσουμε με αυτήν την soft law και το πλαίσιο συνεργασίας και έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για μία οδό, μία κατεύθυνση την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε και στο μέλλον, καθότι βασίζεται στην συνένεση, στη συνεργασία μεταξύ των Υπουργών Παιδείας, βοηθώντας τους στις πολύ χρήσιμες και απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Τώρα θα σας απαντήσω για τον προϋπολογισμό. Υπάρχουν ε, από τη μια μεριά οι εθνικοί προϋπολογισμοί και το μήνυμα της Επιτροπής είναι πάρα πολύ σαφές. Χρειάζονται μέτρα για την ανάκαμψη, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν περικοπές στις μακροχρόνιες επενδύσεις. Όταν περάσει η κρίση, η ανάπτυξη βασίζεται σε αυτού του είδους επενδύσεις. Έρευνα, παιδεία κτλ. Αυτό για τον εθνικό προϋπολογισμό. Τώρα ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν είναι εντυπωσιακός για τους νέους και την παιδεία και τον πολιτισμό, παρόλα αυτά αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσιονομικές πρόπτικες και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μην το εγκαταλείψουμε στο μέλλον. Θέλουμε ή δεν θέλουμε να ενισχύσουμε την κινητικότητα, το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης και πιστεύω ότι αυτή η πρωτοβουλία θα στηριχθεί και από την Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο στο μέλλον. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε με το πρόγραμμα Lifelong Learning, κατάρτιση διαβίου και το πρόγραμμα για, την ε, ευρωπαϊκή, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τώρα, το θέμα του Εράσμους και εάν πρέπει ναι ή όχι το Εράσμους να επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Όντως, το σήμα έρασμος είναι κάτι που αντιμετωπίζεται με πολύ θετικό τρόπο στην Ευρώπη. Οι νέοι ανταποκρίνονται θετικά στο έρασμος και όχι μόνο στους φοιτητές και άλλοι νέοι επαγγελματίες. Το έρασμος οδήγησε σε πολλά λοιπόν θετικά, πολλοί νέοι γνωρίζονται, παντρεύονται, δημιουργούνται νέα δίκτυα ευρωπαϊκά. Υπάρχει και το εράσμους Mundus, πάρα πολύ σημαντικό δίκτυο. Είναι το άνοιγμα της Ευρώπης σε όλο τον κόσμο και σε φοιτητές άλλων υπήρων και άλλων χωρών. Είτε λοιπόν θα ονομαστεί έρασμος, είτε θα ονομαστεί κάπως αλλιώς, θα πρέπει να επεκταθεί. Και όταν μιλάμε παραδείγματος χάρη για εράσμους των ε, ασκούμενων, αυτό είναι ουσιαστικά το το Λεωνάρντο. Αυτό λοιπόν λίγο με ενοχλεί το ότι το ονομάζουμε και αυτό Εράσμους, αλλά εν πάση περιπτώσει όποια και να είναι η ονομασία, σκεφτόμαστε όλο και περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω ότι και εσεί θα το κάνετε, μέχρι που μπορούμε να επεκτείνουμε, αν θέλετε, αυτήν την επιτυχία, η σχετική επιτυχία του προγράμματος Εράσμος. Η κυρία Πακ έτσι μας οδήγησε στο Κομένιους. Ξεκινήσαμε δηλαδή από το Εράσμους και την επιτυχία του και οδηγηθήκαμε στο Κομένιους που είναι για τα σχολεία. Τώρα, θα τα ονομάσουμε όλα Εράσμους ή θα τους δώσουμε άλλο όνομα. Αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει να προωθήσουμε, να ενισχύσουμε την κινητικότητα και όποιο και να είναι το οικονομικό μας, η οικονομική μας βάση και ο προϋπολογισμός θα πρέπει να δούμε να συμμε... πώς μπορούν όλοι να συμμετάσχουν ο κόσμος των επιχειρήσεων, οι τράπεζες, η κεντρική τράπεζα, έτσι ώστε να δώσουμε μια νέα όθηση. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που μπορεί να ενισχυθεί στην διάρκεια της θητείας σας η Επιτροπή Μπαρόζο 2 σίγουρα με τις νέες δημοσιονομικές σας προοπτικές θα θίξει και τα θέματα του πολιτισμού. Η κυρία Ναβολάκοβα έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Στήριξη στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ναι, είναι μία από τις κύριες αποστολές των διαρθρωτικών ταμείων και των κοινωνικών ταμείων. Εγώ ήμουν ε, στην Διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης προηγουμένου και αυτό ακριβώς κάναμε για να στηρίξουμε δημιουργίες θέσεις απασχόλησης σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό όμως δεν είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Φεύγουν Σλοβάκοι φοιτητέ και πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι μόνο. Πολλοί φοιτητέ έρχονται στις νέες χώρες γιατί έχετε αναπτύξει, παραδείγματος χάρη, μαθήματα στα αγγλικά και έτσι προσελκύεται φοιτητέ οι οποίοι έρχονται μη γνωρίζοντας καταρχήν τη γλώσσα της χώρας και κατόπιν την μαθαίνουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να στηρίξουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και η κατάρτιση και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης εδώ συμβαδίζουν. Για το Google. Επεξεργαζόμαστε διάφορες προτάσεις και όσον αφορά την επεξεργασία των βιβλίων, την ψηφιακή αν θέλετε παρουσίαση των βιβλίων μέσω του Google, πιστεύω ότι η συζήτηση ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Το Europeana, το οποίο θα συζητήσετε αύριο και είναι υπεύθυνη η Γενική Διεύθυνση Κατάρτισης, είναι μία πτυχή. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν οι εταιρικέ σχέσεις με τρίτες χώρες, υπάρχει ο ανταγωνισμός, υπάρχει ο πολιτισμός που εκπροσωπώ εγώ, υπάρχει και η κοινωνία της πληροφορικής. Θα πρέπει λοιπόν με ισορροπημένο τρόπο να προσεγγίσουμε το Google, τις δυνατότητες που προσφέρει, αλλά και την προστασία του βιβλίου στην Ευρώπη. Είναι ένα θέμα κλασικό, αν θέλετε, για το πώς θα γίνει το mainstreaming στον πολιτισμό. Η ψηφιακή ατζέντα είναι κάτι που περιέχει πολλά θέματα και αυτό. Όντως λοιπόν το συζητάμε το θέμα αυτό με πολύ πολύ έντονο και ενδιαφέροντα τρόπο και βεβαίως για το θέμα αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να υπάρξει μια θεσμική συζήτηση. Υπάρχει ακόμα μια ερώτηση. Η κυρία Κώστα, συγγνώμη την ξέχασα. Grazie. E σας ευχαριστώ. Εκτίμησε ιδιαίτερη την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας και το σενάριο που μας παρουσιάσατε, κυρία αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω μια πτυχή. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό από στρατηγικής άποψης πλέον η Ευρώπη να μιλά για πολιτιστικές πολιτικές και όχι μόνο για πραγματικότητα. Μιλάμε για, αυτό είναι το μεγάλο βήμα του 2007, το ότι αυτό πλέον αναγνωρίζεται. Και όσον αφορά τον προπολογισμό, όλο αυτό το πολύ σημαντικό σενάριο, αυτή η ενδιαφέρουσα στρατηγική ένταξη των πολιτιστικών πολιτικών σε όλες τις κοινωνικές πολιτικές, το mainstreaming, ε, μα βοηθά να καταλάβουμε τη σημασία αυτή τη προπτικής. Και διαρωτώ σε σχέση με το γεγονό ότι συμμερίζομαι πολλά από τα όσα είπε η κυρία Κέντα, ιδιαίτερα όταν τοποθετεί στο, επίκεντρο της ε,